Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ώρα περνάει. Ξεναρχίζουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των εκτελεστικών οργανισμών που βρίσκονται εδώ για την ανταλλαγή απόψεών μας, όπως συμβαίνει ετησίως, για τον προπολογισμό των οργανισμών. Φέτος, οι οργανισμοί εκπροσωπούνται από τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Επιστημιστική Ασφάλεια, ο οποίος είναι και πρόεδρος του όλου δικτύου. Με την ε, συμφωνία του εισηγητού μας, του μόνιμου εισηγητή μας ε, για τους οργανισμούς του κυρίου Γκάγερ, δίνω αμελητή το λόγο στον κύριο Πιόλ της ΕΦΣΑ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, αγαπητά μέλη. Ευχαριστούμε που καλέσατε το δίκτυο στην ε, συνεδρίασή σας, που είναι σταθερό ραντεβού μας στην ε, όλη διαδικασία προπολογισμού. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία αυτή να παρουσιάσουμε τη δική μας άποψη για τον ε, προπολογισμό. Καταρχάς να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερος το ότι το σχέδιο προπολογισμού του 2018 θα επικεντρωθεί στην ε, ανταγωνιστικότητα, στην ε, μετανάστευση, στις θέσεις εργασίας και οι ε, κατανομές των ποσών έχουν γίνει σύμφωνα με αυτές τις προτεραιότητες. Προφανώς ο δικός μας ο ρόλος ως δικτύου και ως συντονιστών του δικτύου δεν είναι να επικρίνουμε ή να συζητήσουμε τις πολιτικές αποφάσεις για το πώς επενδύονται οι πόροι της Ένωσης. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε οριζόντια θέματα, τα οποία θα επηρεάσουν την αποτελεσματική λειτουργία των 45 υπηρεσιών. Και θέλουμε να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, που επίσης έχουν αναφερθεί από τις επιμέρους ε, υπηρεσίες, από τους επιμέρους εκκληστικούς οργανισμούς, σε επίπεδο γραμματείας. Σύμφωνα λοιπόν με την βασική αυτή θέση και από το 2013 και μετά η βασική μας στόχευση εντός του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι η μείωση του προσωπικού. Το 5 5% δηλαδή και το σχετικό πρόγραμμα μειώσεων που περιγράφεται στο, στην ανακοίνωση της Κομισιόν του Ιουλίου του 2013 και ε, βεβαίω άλλε εξελίξεις που ε, επηρεάζουν την ε, απόδοση των οργανισμών. Αυτό θέλω να πω καταρχάς και Θέλω να πω ότι θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι οι οργανισμοί έχουν κάνει την, το πρώτο 5% των μειώσεων από το 2016. Έγινε λοιπόν αυτό. Και εξεκολουθούμε να είμαστε αναφανδόν αντίθετοι με, την, με, αυτή την, με αυτό το πουλ ανα, μετάθεσης του προσωπικού. Είναι ανεπαρκές και είναι και αναποτελεσματικό. Θεωρώ ότι πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Και για λόγους αποδοτικότητας δηλαδή. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, Ακόμη και αν αυτό το πουλ έχει εφαρμοστεί πλήρως if if και αν ε, υπολογίζουμε και τα νέα καθήκοντα που έχουν δοθεί στους ε, οργανισμούς όπως ας πούμε η ασφάλεια, η μετανάστευση, η οικονομική εποπτεία και τα αντιπαραθέσουμε με το προσωπικό και τις μειώσεις έχουμε ουσιαστικά λάβει και εφαρμόσει ένα 10% των μειώσεων του προσωπικού. Οπότε το 5 5% έχει εφαρμοστεί σχεδόν πλήρως για το 2018. Οπότε χαίρομαι που αναγνωρίζεται και αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την πρότασή της του προπολογισμού και χαιρόμαστε που το Ελεκτικό συνέδριο επίσης κάνει μια πλήρη αξιολόγηση αυτού του περίπλοκου θέματος για να δώσουμε περισσότερο φως στο πώς έχει εξελιχθεί το προσωπικό των οργανισμών τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια αυτή τη ε, προσέγγιση εντός του προπολογισμού. Οι μειώσει του προσωπικού είναι ένα σημαντικό συγκεκριμένο πρόβλημα για την πλήρη λειτουργία των ε, υπηρεσιών, των οργανισμών, που σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση της αναδιάταξης ε, ξεπερνούν τις, ε, τους περιορισμούς και τις μειώσεις του προσωπικού ε, σε σχέση με, άλλους, με άλλα θεσμικά όργανα. Και αυτό μεγεθύνεται αν δείτε ότι όταν ε, λειτουργούν πλήρως οι ε, υπηρεσίες έχουν ήδη υποβάλει μέσω της, των αποφάσεων των διοικητικών του συμβουλίων ε, αιτήσει για επιπλέον προσωπικό λόγω του αύξηση του φόρτου εργασίας. Και αν αυτό το προσμετρήσετε, ακριβώς λόγω του νέου φόρτου εργασίας, με, ναι, και τις αρνητικές απαντήσεις βεβαίως που έχουμε λάβει, αλλά και τις μειώσεις του προσωπικού, βλέπουμε ότι καταλήγουμε σε μια προσέγγιση διατήρησης του προσωπικού σε ένα 20% για, την, για τις υπηρεσίες που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά επηρεάζεται η λειτουργία, η αποδοτικότητα των εκτελεστικών οργανισμών. Και επίσης ε, αναγνωρίζεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο του προπολογισμού 2018 ότι σε κάποιους τομείς όπως η δημοσία υγεία και το περιβάλλον, η απασχόληση και η νεότητα, η νεολαία, οι δυνατότητες των υπηρεσιών να κάνουν τις, ε, τα καθήκοντά τους έχουν επηρεαστεί ακριβώς λόγω αυτής της μείωσης του 10% συν τον, ε, ε, του έξτρα φόρτου εργασία, δηλαδή μείον 20% των δυνατοτήτων των ε, οργανισμών. Οπότε χαιρόμαστε που ο Επίτροπο Ότιγκερ, όταν παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού 2018, δήλωσε ότι οι μειώσει του, του προσωπικού δεν θα πρέπει να προχωρήσουν και μετά το 2019, αλλά θα πρέπει, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσουν κιόλα πριν το 2018. Και συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτό το, αυτή η προσέγγιση αναδιάταξης θα πρέπει να σταματήσει γιατί δεν αιτιολογείται, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι οι υπηρεσίες ε, δεν αισθάνονται μόνο την πίεση λόγω των μειώσεων του προπολογισμού, αλλά και λόγω του έξτρα κόστους και άχθους που έχει να κάνει με την εφαρμογή του οδικού χάρτη της Κομισιόν, όπως ας πούμε έχει το, τα έγγραφα και το single programming, τις αξιολογήσεις, ε, την εξωτερήκευση των ε, ελέγχων από το ελεκτικό συνέδριο και κυρίως ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, αλλά και οικονομικούς και κανόνες για το προσωπικό, που είναι πραγματικά άτεγκτοι, αδικαιολογήτως άτεγκτοι για τη διαχείριση των υπηρεσιών, των οργανισμών αυτών, που είναι ούτως ή άλλως και σε καθήκοντα, αλλά και σε μέγεθος τελείως διαφορετική σε σχέση με τα θεσμικά όργανα. Βλέποντα λοιπόν αυτού του ε, περιορισμού για τον προπολογισμό και βλέποντα και τι ε, μειώσει του προσωπικού, αυτό που έκαναν οι υπηρεσίε ήταν να ενισχύσουν τι προσπάθειε του για να είναι πιο αποδοτικέ και επιμέρου, αλλά και συλλογικά εισάγοντας κοινέ υπηρεσίες και κοινέ προσπάθειες απόδοσης συμβάσεων και θεωρούμε ότι έχουν αποδώσει καρπούς αυτές οι προσπάθειες και έχουν οδηγήσει σε εξοικονομήσεις και σε ό,τι αφορά το προσωπικό αλλά και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και όρια σε αυτή την αποδοτικότητα. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον τα όρια αυτά. κυρίως ε, όταν βλέπουμε τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν οι ε, οργανισμοί. Είναι τόσο άτεντοι και είναι τόσο ε, πολλές οι διοικητικές απαιτήσεις και οι προσπάθειες για την απλούστευση και για την εκλογήκευση των πραγμάτων δεν έχουν δώσει απτά αποτελέσματα. Οπότε θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα θεσμικά όργανα να ξανασκεφτούν και υπό το φως του κανονισμού για το δημοσιονομικό πλαίσιο το κατά πόσο θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε μια προσέγγιση του προϋπολογισμού σε σχέση με την απόδοση. Οπότε να επικεντρωθούμε στην απόδοση και στα αποτελέσματα. Αλλά από την άλλη να δώσουμε και στις υπηρεσίες την ευελιξία που χρειάζονται για να χρησιμοποιούν τους πόρους που έχουν, είτε είναι ανθρώπινοι πόροι, είτε είναι οικονομικοί πόροι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τα αποτελέσματα που έχουμε υποσχεθεί να δώσουμε για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και αν μου επιτρέπετε, δύο λόγια ακόμη για τον ιστορικό συντονισμό και το, την, υπηρεσία, κοινής, την κοινή υπηρεσία υποστήριξης. νομίζω ότι όλοι βλέπετε ότι έχουμε, υπάρχει ενισχυμένος ρόλος ε, εντός, για τον συντονισμό των ε, υπηρεσιών και νομίζω ότι αυτό βοήθησε ιδιαίτερα σε τη φορά την εφαρμογή του οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, την, ε, και τα εργαλεία που υπάρχουν για το σχεδιασμό, για τις απαλλαγές, για τον προπολογισμό κτλ. Και μάλιστα το Κοινοβούλιο πρόσφατα συνέστησε ότι ή το δίκτυο των ε, οργανισμών θα πρέπει να ε, επεκτείνει τη γραμματεία του στις Βρυξέλλες ακριβώς για να διευκολύνει και να εξασφαλίσει αυτές τις ε, δυνατότητες και τον, για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου άχθου εργασίας. Και μάλιστα βοηθά και τις υπηρεσίες, η γραμματεία αυτή και τα θεσμικά όργανα. Δώσαμε λοιπόν μια συνέχεια σε όλα αυτά τα στοιχεία και μετά τη σύσταση του, του Κοινοβουλίου ζητώντα μια ακόμη θέση για, την, ε, για το συντονισμό στα πλαίσια του προπολογισμού 2018 και θα ζητούσαμε να επανεπιβεβαιώσει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στήριξή του στο πλαίσιο αυτό. Αν δούμε τώρα πέραν του 2018, καλωσορίζουμε τη δουλειά που έχει γίνει ε, από την ε, Διαθεσμική ε, Ομάδα εργασία 2. Για μα είναι σημαντικό να έχουμε μοντέλα ε, συνολικά για την κατανομή των πόρων και να έχουμε ευέλικτη προσέγγιση ό,τι αφορά την απόδοση. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τι ευρωπαϊκέ αρχέ του προπολογισμού να ενισχύσουν τι προσπάθειέ του έτσι ώστε να έχουν μεθοδολογίε κατανομή του προπολογισμού σύμφωνα με την απόδοση. Εμεί ω υπηρεσίε επενδύουμε σημαντικά έτσι ώστε να έχουμε μοντέλα που να μπορούν να εφαρμοστούν για όλε τι υπηρεσίε ανάλογα με ένα μοντέλο οριμότητα και μια λογική παρέμβαση που έχει ως ε, στόχο να μπει σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και να δοκιμαστεί από κοινού με όλα τα θεσμικά όργανα. Οπότε εμεί σα λέμε να χρησιμοποιήσετε τους ε, οργανισμούς αυτούς για να δείτε νέους τρόπους ε, κατανομής του προπολογισμού αλλά και ελέγχου αυτού. Θεωρώ ότι θα είναι πιο εύκολο να το κάνετε μέσω των υπηρεσιών και όχι μέσω των μεγάλων θεσμικών οργάνων όπω το Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν. Και επίσης θα θέλαμε να ε, καλέσουμε τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προπολογισμού να εξετάσουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν επιπλέον τρόπους χρηματοδότησης των ε, οργανισμών όπως ας πούμε τα τέλη ή το κόστος ε, προς τους εθνικούς, τις εθνικές διοικητικές αρχές για τις διάφορες δραστηριότητε. Υπό το φως λοιπόν όλων αυτών των εξελίξεων και των προκλήσεων, εμείς ως οργανισμοί θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και την κοινή δουλειά που κάνουμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με βάση βεβαίως την διαφάνεια. Ελπίζω ότι αυτό μπορείτε να το δείτε. Οι υπηρεσίε ε, αυξάνουν και τη δική τους διαθεσιμότητα να είναι απολύτως διαφανής και βεβαίω να, να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και βεβαίω θα θέλαμε να ξαναέρθουμε εδώ έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε τα αποτελέσματα ω εταίροι στις διάφορες διαδικασίε που τρέχουν, όπως ας πούμε η ολοκλήρωση της δουλειά για την διαθεσμική ομάδα εργασία, το Brexit, τα σχέδια για το 2020 κτλ. Σα ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστω να απαντήσω στι ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσίασή του, η οποία φέρνει στην επιφάνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εξωτερικές αυτές τις υπηρεσίες λόγω της μείωσης του προσωπικού. Κάποιες προτάσεις τις οποίες κάνετε έτσι ώστε να υπάρξουν συμπληρωματικοί πόροι για τις ε, εξωτερικές αυτές υπηρεσίες που δεν θα είχαν συνέπεια την αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής μας τώρα, ο κύριος Γκάιερ, πώς βλέπετε τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάλι βρισκόμαστε σε μια κλασική περίπτωση για το πώς μεταχειρίζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τους ε, του οργανισμού. Δύο αλλάζουν έδρα από το Λονδίνο ε, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Υπηρεσία ε, και άλλη μία υπηρεσία πρέπει να αλλάξουν έδρα και βεβαίω συμβαίνει πάντα αυτό που συμβαίνει συνήθω. Κάποιες, ε, η μία εκ των δύο ε, έχει πολλές περισσότερες ε, προσφορές για μεταφορά της έδρας της για την, και νομίζω ότι και η άλλη θα έχει αρκετές προσφορές. Πάλι βρισκόμαστε λοιπόν σε μια παρόμοια κατάσταση όταν πρόκειται για μετάθεση των εδρών των υπηρεσιών. Τότε, όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, τα κράτη-μέλη μπαίνουν σε μια διελκυστίνδα, σε, μια, σε έναν ανταγωνισμό δυνάμεων για το πού θα καταλήξουν τελικά αυτές οι υπηρεσίες. Ε, θυμόμαστε τι έκανε και ο Μπερλουσκόνη με την, ε, όταν πήρε την ΕΦΣΑ και την πήγε στην Πάρμα. Αλλά βεβαίως ε, μετά οι υπηρεσίε αυτές γίνονται πραγματικά πάρα πολύ δαπανηρές. Έχω πει πολλές φορές... έχω βρίσκονται οι υπηρεσίες αυτές ε, σε μια κατάσταση όπου ε, όπως ένα ε, μπάσταρδο παιδί του μεσαίωνα μεγαλώνει με αγάπη μένα, αλλά καμιά φορά βρίσκεται και λίγο στη μέση όλων χωρίς να ξέρει κανείς τι να το κάνει. Εμένα επειδή έχω σπουδάσει ιστορία πάντα με ενδιέφεραν τέτοιου είδους συγκρίσεις. Οπότε τώρα θα, βρω, θα βρεθούμε στην εξή κατάσταση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιπαρατεθούν το ένα με το άλλο. Και το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες βεβαίως μπορεί να, είναι, μπορεί να καταλήξει σε κάποιο ε, αποτέλεσμα. Ήταν ούτως ή άλλως, ε, παλιά απόφαση για την ρυθμίση της ε, αγοράς ε, να μοιραστούν σε τρεις διαφορετικές πόλεις οι τρεις αντίστοιχες υπηρεσίες, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Φραγκφούρτη ας πούμε. Και Νομίζω ότι στο τέλος η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Υπηρεσία δεν θα ενσωματωθεί με, άλλες, με τις άλλες δύο ήδη υπάρχουσες. Μάλλον θα την, θα τη βρούμε σε μια άλλη ωραία πρωτεύουσα της Ευρώπης, γιατί έτσι θέλει το Συμβούλιο. Τέτοιες καταστάσεις όμως πρέπει να τις έχουμε πάντα υπόψη, κυρίως όταν βλέπουμε και τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό. όταν ανταλλάσσουμε επιχειρήματα για το τι κάνουμε με τις υπηρεσίες και πώς μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Νομίζω ότι ε, αυτό το πουλ της αναδιάταξης είναι πραγματικά πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Ήταν λίγο περίπλοκη η ιδέα. Συμμερίζομαι την άποψη δηλαδή των υπηρεσιών και συμμερίζομαι και την άποψη ότι το ιστορικό ήταν αυτή η συμφωνία του 5% μείωσης με, σύμφωνα και με το ενδιάμεσο σχέδιο ε, του πολιετούς πλαισίου. Ίσως να μην χρειαζόταν κατά ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο και ταυτόχρονα η απόφαση ήταν ότι ήταν, είναι σημαντική και απαραίτητη η ανάπτυξη, η εξέλιξη των ε, υπηρεσιών γιατί όντως ε, προκύπτει πάρα πολύ περισσότερος φόρτος εργασίας. Κάτι που έπρεπε να γίνει μέσω αυτού του πουλ, μέσω αυτής της αναδιάταξης. Και ο Γενικός Διευθυντής μίλησε ακριβώς για αυτό το 5% των μειώσεων στο προσωπικό. Τα προηγούμενα χρόνια, όντως, βέβαια, κάποιες υπηρεσίες δεν ήρθησαν στο, στο ύψος των υποχρεώσεών τους. Τώρα κάποιες ε, εθνικές ε, αντιπροσωπείες ε, εκπλήσονται όταν λένε ότι δεν έχουμε δεύτερη ομάδα μεταφραστών για την συνεδρίασή σας. Ίσως λοιπόν και σε αυτή την κατάσταση να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να μειώνουμε συνέχεια το προσωπικό και να περιμένουμε μονίμως το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό αυτό να είναι στο ίδιο επίπεδο. Εγώ μίλησα με τον Επίτροπο Ετινιέρ και θα ήθελα και οι ε, συνάδελφοι να το προσέξουν. Το 2018 είναι το τελευταίο έτος αυτής της προσέγγισης αναδιάταξης. Θα έχουν τελειώσει μετά τα πέντε χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα δεν θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Οπότε ως προς αυτό μπορούμε ίσως κάποια πράγματα να διορθώσουμε, να δώσουμε για κάποια συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, χρήματα επιπλέον στις υπηρεσίες. Θα πρέπει να δούμε ποιες επιλογές έχουμε και υποστηρίζω και την πρόταση να σκεφτούμε πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Σε λίγες μέρες θα μιλήσουμε για την αναδιατύπωση του κανονισμού για την ΕΣΑ. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε για το ότι μια υπηρεσία που ε, ε, προσφέρει υπηρεσίες δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη. Φυσικά μπορεί. Οπότε θα πρέπει να προσφέρουν μια τέτοια δυνατότητα στις, σε κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στο παρελθόν το είχα πει, είχα προσπαθήσει να το πω, γιατί κάποιες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει, υπάρχει τρίτη ομάδα, είτε η ΕΣΑ, είτε η βιομηχανία, που πληρώνει τέλη, η Κομισιόν και οι αρχές προπολογισμού δεν θα πρέπει να μπορούν να τις διαγράψουν, γιατί ουσιαστικά ε, καταβάλλονται τέλη. Οπότε είναι οι υπηρεσίες οι οποίες ε, αποδίδονται σε τρίτους από τις υπηρεσίες μέσω καταβολής τελών. Άρα έτσι υπάρχει μια ε, χρηματοδότηση ουσιαστικά των υπηρεσιών αυτών και νομίζω ότι αυτό είναι μια λογική λύση. Ανησυχώ βεβαίω ελαφρώ για το τι θα γίνει με αυτό που είπατε εσείς κύριε Διευθυντά για το πώς μπορεί να μετρηθεί η απόδοση, η αποδοτικότητα των υπηρεσιών. Υπήρχε μια τέτοια προσέγγιση, την ξεκίνησε η Κομισιόν ε, με την ΕΑΣΑ στην Κολονία, την παρακολουθούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αλλά με τους τριμερείς ε, διαλόγους με το Συμβούλιο πάντα βρισκόμαστε, αντιμετωπίζουμε τεράστια άρνηση. Δεν ξέρω, είναι ξεροκέφαλα τα κράτη-μέλη, δεν ξέρω. Μια, ένα σκόπιμο, εν πάση περιπτώσει, εύλογο επιχείρημα ακόμη δεν έχω ακούσει. Συζητούμε πάντα για την προσέγγιση της ε, Επιτρόπου Γεωργίευα για το budgeting on results, ε, κατανομή του προπολογισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα και γιατί να μην το σκεφτούμε αυτό να ισχύει και για τις υπηρεσίες που έχουν καλή απόδοση. Με βάση λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να, το... να, λύσουμε το πρόβλημα με το αδιέξοδο που μας φέρνει πάντα το Συμβούλιο. Εγώ θέλω να βοηθήσω και χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Χαίρομαι που βρήκατε το δρόμο προς το Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση για, τις, για το μέλλον των υπηρεσιών. Ξεκινάει η συζήτηση για τους συναδέλφους που το επιθυμούν. Α, συμφωνούμε όλοι. Πάντως έχουμε την αίσθηση από χρόνο σε χρόνο ότι επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε τα λόγια μας να οδηγήσουν σε δράσεις. Η ομάδα Μόντι δεν ασχολήθηκε με τους ιδίους πόρους για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορεί να χρεώνουν τις υπηρεσίες τους, τα τέλη τους, τα ρόγελτη τους. Πάντως ε, το θέμα είναι να βρούμε κάποιο τρόπο δημοσιονομικά για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές και μερικές φορές βλέπουμε να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στις ευρωπαϊκές αυτές εξωτερικές υπηρεσίες και τις αντίστοιχες εθνικές. Θα ξεφύγουμε ποτέ από τους εθνικούς εγωισμούς. Αν όχι τα πράγματα θα πάνε άσχημα. Και βλέπω επίσης ότι υπάρχουν πολλές, πιο, πολλές υποψήφιες πόλεις για να υποδεχθούν τις εξωτερικές υπηρεσίες παρά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κυρία Τωμά έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως να διαφωνήσω λίγο με αυτά που είπατε. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι τα τέλη η τιμή των υπηρεσιών που παρέχουν είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Το είδα αυτό πως λειτουργεί το σύστημα στις εθνικές υπηρεσίες. Είδα τι συνέπειες έχει κάτι τέτοιο. Από τη μία βλέπω τις υπηρεσίες αυτές να αλλάζουν τις αποστολές τους και να ασχολούνται με θέματα τα οποία είναι προσοδοφόρα και να εγκαταλείπουν τις αποστολές οι οποίες δεν, ε, δεν αποδίδουν χρήμα. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει επίσης εξάλλου και σε συγκρούσεις συμφερόντων και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε έτσι εύκολα. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική λοιπόν και θα ήθελα να είμαι βέβαιη ότι ούτε αποστολή, αλλαγή αποστολής θα υπάρξει ούτε ε, σύγκρουση συμφερόντων. Τότε μόνο θα συμφωνήσω. Κοιτάξτε, το επειδή ε, δεν υπάρχουν τέλη δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, αλλά υπάρχει κανένας λόγος να αυξήσουμε τους κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι οι οργανισμοί θα έπρεπε να έχουν άλλη προβολή στη δουλειά που κάνουν για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί κάποιοι, ε, πολιτικοί, πολιτικοί θύνοντες συνειδητοποιούν την ύπαρξη των οργανισμών μόνο όταν αποφασίζεται ότι μπορεί να αλλάξει η έδρα τους, όπως έγινε με τον Brexit. Οπότε η προβολή των οργανισμών είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι προς όφελος και των ίδιων των οργανισμών. Κατά δεύτερον, η αναδιάταξη στους δύο οργανισμούς η ύπαρξή τους η ίδια, που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να μετατραπεί, σημαίνει ότι θα συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή με τον γεωγραφικό τους εντοπισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, ισότιμη κατανομή γεωγραφικά. Δεν έχει νόημα στην ίδια πόλη να συγκεντρώνονται πάνω από δύο οργανισμοί. Κατά τρίτον, για το θέμα των περικοπών και ως προς τις αρμοδιότητες και την ε, αντίφαση που μπορεί να υπάρχει. Από τη μια να απαιτούμε περικοπές, 5% στο προσωπικό, το staff, και από την άλλη από άλλους οργανισμούς να απαιτούμε περισσότερες ε, αρμοδιότητες που πρέπει να φέρουν εις πέρας. Το ερώτημα είναι, εάν αυτές οι περικοπές για μείωση των δαπανών συνδυάζονται και με κόστος, διότι το, δε, το ότι δεν πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις πολλές φορές μεταφράζεται σε κόστος. Το ότι δεν δεν εφαρμόζονται ε, κάποιες ενέργειες σε συγκεκριμένους χώρους, έχει κόστος πολλές φορές. Κόστο μεγαλύτερο από ότι αυτά που εξοικονομούνται. Είναι λοιπόν σημαντικό να σημειώσουμε ε, τι αντίκτυπο, τι κοινωνικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν ε, αυτές οι περικοπές του 5%. Το άλλο ερώτημα και σε σχέση με, το, με την κατάρτιση προπολογισμού βάσει των επιδόσεων. Ανέκαθεν λέγαμε ότι είναι κάπως δύσκολο να εφαρμοστεί στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως το ερώτημα είναι εάν ο στόχος αυτός Η ανάγκη αυτή να υπάρξει προσανατολισμό προ ε, αποτελέσματα, επιδόσεις, εάν έχει διαπιστωθεί και στου οργανισμού και αν κατά κάποιο τρόπο έχει εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι σημαντικό είναι ο συντονισμό και με του εθνικού φορεί, με του εθνικού οργανισμού. Είναι σημαντικό να είναι καλό ο συντονισμό. Πέραν αυτού όμω, ο συντονισμό είναι κάτι το δεδομένο που πρέπει να υπάρχει. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ποιος άλλο θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω απολύτω με τον κύριο Φερνάντε και με εσά, Πρόεδρε, με όσα είπατε. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σα. Γνωρίζω ότι έχουμε αυτή την δυσκολία, ότι δημιουργούμε οργανισμού και μετά έχουμε προπολογισμού που μικραίνουν όλο ένα. Ιδίω μετά το 2020 θα μικραίνουν κι άλλο. Θα πρέπει όμω να καλύπτουμε όλα τα απαραίτητα κόστη. Διότι έχουμε αυτή τη διαρκή μείωση του προσωπικού και τότε καταλήγουμε στο ερώτημα χρειαζόμαστε πραγματικά τους οργανισμούς και αν ναι ποιους. Δύο απαντήσεις λοιπόν είναι λογικές. Είτε βρίσκουμε άλλη πηγή χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, διότι δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά αυτή η διαφορετική πηγή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβληθεί επιπλέον άχθο στι επιχειρηματίε, εταιρείε και πολίτε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτό το επιπλέον βάρος. Αλλά μπορούμε να τους ρωτήσουμε τους ίδιους ε, και να απευθυνθούμε σε αυτούς. Εταιρείε που μπορεί να έχουν συγκεκριμένες σχέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς. Να τους ρωτήσουμε αν αισθάνονται ότι χρειάζονται αυτόν τον οργανισμό. Τους αποκομίζει ωφέλη. Διότι τότε μπορεί να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον τέλη για να ε, συνεχίσει να υπάρχει οργανισμός. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί να μην το προβλέψουμε εάν συμφωνούν αλλά να μην το επιβάλλουμε, μην επιβάλλουμε πλέον τέλη. Δεν θα ήταν εύστοχο. Ε, η προσέγγιση bottom-up, από κάτω προς τα πάνω, εδώ θα μπορούσε να είναι εύστοχη. Και κατά τα άλλα πρέπει να σκεφτούμε και το εξή. Υπάρχει ίσως δυνατότητα να συγχωνευτούν κάποιοι οργανισμοί για να υπάρχει οριζόντια διοργάνωση και το οριζόντιο κόστος λειτουργίας. Και έτσι βλέπουμε πώς θα του οργανώσουμε διαφορετικά. να σας επισημάνω ότι είχαμε μια απορία και για έναν οργανισμό που είναι στην Ελλάδα. Σε δύο διαφορετικά σημεία, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Άλλαξε αυτό, ε, έγινε κάτι ή ε, λήφθη κάποια απόφαση ή κάθε χρόνο θα καταλήγουμε στην ίδια διαπίστωση. Ήσουν λοιπόν υπό τη δική μας ε, αρμοδιότητα και ευθύνη να πιέζουμε για να γίνουν αλλαγέ και να ε, εντοπίζουμε ποιοι είναι οι οργανισμοί που μπορούν να συμβάλλουν λόγω χάρη στην ασφαλή της αεροπλοείας. Οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν γοργά και αυτό ωφελεί και τους κατασκευαστές αεροσκαφών. Υπό αυτές τις συνθήκες λογικό είναι να, να χρηματοδοτήσουν, να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση των οργανισμών οι κατασκευαστές λόγω χάρη. Κύριε Γκάγερ, Κάτι είπατε και εσείς για τους δύο οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια. Για την εκπαίδευση των αστυνομικών, ε? Πώς έχει προχωρήσει αυτό. Äh, Καλή ερώτηση. Ε, θα τη ρωτήσω και εγώ στο Συμβούλιο με τη σειρά μου, Πρόεδρε. Χωρίς τώρα να θέλω να επικρίνω βεβαίως τους αξιότιμους συναδέλφους. Εδώ κάνουμε την ίδια συζήτηση και για 10, και 10 λεπτά λέμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ότι θέλουμε οργανισμούς και από την άλλη θέλουμε να υπάρξουν και συγχωνεύσεις αν γίνεται. Έχουμε λοιπόν δύο καταστάσεις όπου οι υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δύο έδρες. Και καμιά φορά τα κράτη-μέλη αποφασίζουν πού θα είναι η έδρα στην επικράτειά τους. Ας πούμε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων έχει έδρα στην Βαλενσιάν και έχουν και τα κεντρικά τους στη Λίλ. Έτσι ώστε οι επισκέπτες με το ΤΕΖΕΒΕ, το τρένο, να μην χρειάζεται να κάνουν και το ταξίδι από τον σταθμό μέχρι το Βαλενσιέν. Ε, τώρα, πόσο ε, ε, έξυπνο είναι αυτό, πόσο σωστό να έχουμε σε τόσο απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης υπηρεσίες, πρέπει να το δούμε. Και το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στην Ελλάδα. Έχει την έδρα της στο Ηράκλειο, αλλά επειδή κανένας δεν θέλει να δουλέψει εκεί, γιατί δύσκολα φτάνει κανείς στο Ηράκλειο σε σχέση με την Αθήνα, υπάρχει και η έδρα στην Αθήνα. Δεν προετοιμάστηκα για το πόσο έχουν προχωρήσει τα πράγματα εκεί, αλλά για την Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά ο Γενικό Διευθυντή ήταν ε, πολύ αισιόδοξο ότι είχαν φτάσει σε μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Ότι να πάει δηλαδή πλήρω η έδρα τη υπηρεσία στην Αθήνα. Και όλοι όσοι ε, είπανε ότι ναι, αλλά θέλουμε δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες υπηρεσίες, ανεξάρτητα για το, τι είναι, για το ποιο πράγμα είναι υπεύθυνε, θα πρέπει να φτάσουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης. Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν υπηρεσίες, αλλά μπορεί να βρεθούμε και μπροστά σε καταστάσεις όπου το λογικό θα είναι για την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, ας πούμε, που βρίσκεται όταν σε μια απομακρυσμένη περιοχή στον Ηνωμένο Βασίλειο, να μην κάνουν την αλλαγή μαζί με τις άλλες υπηρεσίες για την ε, δικαστική και την αστυνομική συνεργασία και όπου θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες και συνεργασία καλύτερη και που θα μπορούσαν ίσως να, πούνε, να, να, να Όχι, αυτή η υπηρεσία βρίσκεται στη Βουδαπέστη. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσε κανείς να σας πει και πέντε επιχειρήματα γιατί είναι μάλιστα το σωστό σημείο να η Βουδαπέστη για αυτή την υπηρεσία. Γιατί μόνο η Ουγγαρία ξέρει καλά τα αστυνομικά θέματα από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει να θυμίσω και τη συζήτηση που κάναμε χθες για άλλα θέματα δεν μπορούμε δύο πράγματα να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να λέμε το Ζάγκρε πρέπει να έχει την επόμενη υπηρεσία γιατί είναι δίκαιο, το κράτο μέλο αυτό να έχει, να έχει μια υπηρεσία και ταυτόχρονα να λέμε ναι, αλλά θα μπορούσαμε ίσω να έχουμε και έδρα. Ε, Ευτυχώ, ε, συσσαγωγικά, αυτό έχει μείνει στα χέρια του Συμβουλίου και έχουμε τις, ε, έχουν γίνει ήδη κάποιες προσφορές για τις έδρες των υπηρεσιών. Νομίζω ότι δεν έχουμε προσανατολιστεί στην απόδοση των υπηρεσιών ως προς την επιλογή της έδρας τους. Και μάλιστα κάποιες υπηρεσίες λένε εμείς πρέπει να υπάρχουμε για πάντα. Αν τα καθήκοντά τους μπορούν να γίνουν καλύτερα ή να αναλυφθούν καλύτερα, δεν υπάρχει πρόβλημα να συγχωνευτούν ε, οι υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι χάνεται η έδρα τους. Και μετά και ο, ο δικός μας ο οίκο φέρεται εγωιστικά. Θέλουμε κατευθυντήρες γραμμές για όλες τις υπηρεσίες για την πολιτική απασχόληση. Εγώ ζήτησα, συζήτησα με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης για το αν είδανε το θέμα των ε, συνεργειών μεταξύ υπηρεσιών. Απάντηση εξ όλων, ε, ας μην πιέζουμε τις υπηρεσίες. Πολύ στενή είναι η συνεργασία των υπηρεσιών όταν γίνεται, αλλά αυτό είναι καλό μεν για τις υπηρεσίες, αλλά βεβαίως όταν υπάρχει καλή συνεργασία αυτό είναι κοπλιμέντο για τις υπηρεσίες, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μειωμένη πρόσβαση σε θέματα συγχώνευσης. Και τέλος, για το θέμα των τελών. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλούμε σε λιγότερο ιδεολογική βάση. Τα τέλη, τουλάχιστον για το δικό μας το κράτος, τα διοικητικά τέλη, σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα και τις δημόσιες υπηρεσίες, προφανώς ε, υπάρχουν. Όταν κάποιο θέλει να παντρευτεί, ας πούμε, ε, προφανώς πρώτα πρέπει να πληρώσει. Εμείς δεν αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί ισχύει αυτό. Ε, και όταν συζήτησαμε τη βιομηχανία, δεν μου είπαν ότι δεν είναι δυνατόν. Μου είπαν τι θα πάρω εγώ για τις υπηρεσίες που προσφέρω. Και η υπηρεσία για, τη, για τις αερομεταφορές μου είπαν ότι αν τα δικά μας τέλη ουσιαστικά βελτιώνουν τις υπηρεσίες της ΕΑΣΑ και μπορούμε να έχουμε εμείς καλύτερες ε, επιστοποιήσεις και πιο γρήγορες διαδικασίες, ευχαρίστως να τα πληρώσουμε τα λεφτά. Οπότε δεν χρειάζεται να λέμε Εντάξει, εγώ είμαι... Ε, οι σοσιαλιστέ μιλάνε για το ότι πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από τη βιομηχανία. Εγώ είμαι διαφορετικού άποψη, αλλά το θέμα ουσιαστικά είναι τι θα πάρουμε τελικά. Τι θα πάρει η βιομηχανία για αυτά τα, τέλη. Αυτό θα αποφασίσει το κατά πόσο θα δεχθούν να δώσουν τα τέλη. Και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό στις, ε, στους οργανισμούς για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτή είναι καλή η θέση. Η Ιζαμπέλ δεν έχει άδικο κατά ανάγκη. Υπάρχουν και άλλες σημαντικέ υπηρεσίε ε, σημαντικές υπηρεσίες από τους οργανισμούς και βεβαίως πρέπει τα θέματα σύγκρουση συμφερόντων να τα έχουμε υπόψη μας, αλλά νομίζω ότι ε, έχουμε αρκετά καλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, οπότε δεν ανησυχώ πολύ. Και στο, και στο τέλος αυτό είναι το θέμα που πρέπει να αποφασίσει η ε, Επιτροπή μα. Αν μπορούμε να έχουμε απαλλαγή του προπολογισμού και αν αυτό μπορεί να γίνει μέσω τη επιβελή τελών, γιατί όχι. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα γίνουν πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει στη σοσιαλιστική ομάδα για τα τέλη αυτά. Ο κύριος Φερνάνδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ε, ανάλυση που μόλις έγινε. Η αρχή της μη συγκέντρωσης είναι μια αρχή σημαντική. Η αρχή της μη συγκέντρωσης γεωγραφικός ευνοεί την εδαφική συνοχή. Είναι μια καλή αρχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται. Εάν θέλουμε να ε, συγκεντρώνουμε τα πάντα με το επιχείρημα ότι έτσι κι εκεί όλα γίνονται, ε, με συγχωρείτε, αλλά να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική θα πρέπει όλες, όλοι οι οργανισμοί να έρθουν στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρνατε να το περάσετε αυτό, αλλά τι να πούμε. Ε, εδώ έχουμε όλα τα μέσα συγκοινωνίας. Ε, η λογική είναι εδώ τα έχουμε όλα, οπότε ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ας έρθει εδώ. Ας έρθει ο Μάριο Ντράγκη, ο οποίος επισκέπτεται το κοινοβούλιο. Πώς θα το προασπιστείτε αυτό. Πείτε το στη Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πάει στις Βεξέλλες. Διότι έτσι θα συγκεντρώσουμε εδώ όλους τους οργανισμούς, όλα τα θεσμικά όργανα. Το θέτω ε, και το πάω στα άκρα για να φανεί ότι η λογική αυτή ότι οι άνθρωποι πρέπει να μεταφέρονται γιατί δεν υπάρχει ΤΖΒ. Ε, εντάξει όμως, εάν ε, τα συγκεντρώσουμε όλα σε ένα μέρος, όλα εκεί θα γίνονται. Στη Βιλαβέρδε, στην Πορτογαλία. Ας τα πάμε όλα εκεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, το, το, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν θα χρειάζεται κανένα τεζεβέ. Θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο. Ε, έτσι λοιπόν, επειδή όλοι είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο μέρο, το να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε και τα πάντα δεν έχει λογική. Ε, ο οργανισμό για, το, για, για του σιδηροδρόμου στη Λίλ και στι Βαλανσιέν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει γεωγραφική ε, μη, έλλειψη ισορροπίας και πρέπει να βρούμε την εξισορρόπηση. Αλλά ε, η αρχή τη ενταφικής συνοχή, η αρχή της γεωγραφική ε, είναι αρχές τις οποίες πρέπει να συνεχίσουμε να προσπιζόμαστε. Αυτό που βρίσκω θετικό είναι ότι η συζήτηση θέλει λίγο χρόνο για να πάρει μπρος Νομίζω ότι φτάσαμε ήδη σε ένα ενδιαφέρον επίπεδο. Η κυρία Τωμά. Και εγώ δεν έχω, θα έλεγα, είμαι λίγο θυμωμένη σήμερα το πρωί. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα έλεγα ξεπερνούν τις πολιτικές ομάδες και πολλές φορές οφείλονται απλά ε, στα θέματα γεωγραφικών διαφορών. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια της Ευρώπης σε μια πολύ συγκεντρωτική χώρα. Και γνωρίζω το τι κοστίζει η υπερσυγκέντρωση μέσω της εγκατάλειψης ορισμένων εδαφών. Ο Γένς έρχεται από μια χώρα που δεν είναι συγκεντρωτική και δεν γνωρίζει αυτού του είδους τις ε, υπερβολές εμείς προσπαθούμε εδώ να υπολογίσουμε το κόστος σε επίπεδο θα έλεγα ανεκδοτολογικό της μετακίνησης των υπηρεσιών αλλά δεν υπολογίζουμε το κόστος της έλλειψης της εδαφικής συνοχής και της εγκατάλειψης πολλών περιφερειών. Ο Χωσέ Μανουέλ το είπε, υπάρχει μια βασική αρχή, η αρχή της ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής. Πρόκειται για μία αρχή την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε και για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Από την άλλη, και αναφέρθηκε ο Γένς σε αυτό, υπάρχει θέμα καταλληλότητας για την βέλτιστη απόδοση, δηλαδή να βρούμε περιφέρειες οι οποίες να είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες αποστολές. Αλλά πάντως το να υπάρχει μια σωστή κατανομή είναι βασικό, γιατί αλλιώς θα τα μαζέψουμε όλα εδώ στις Βρυξέλλες. Απ' την άλλη η μισθή είναι πολύ ψηλή στις Βρυξέλλες, λέει ο Πρόεδρος, ενώ στις διάφορες άλλες χώρες είναι πιο φτηνά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες το κόστος της ζωής δεν είναι αυτό των Βρυξελών, οπότε το παράδειγμα δεν είναι το σωστό. Εν πάση περιπτώσει, στο θέμα των τελών, η θέση μου δεν είναι μια ιδεολογική προέλευσης θέση, είναι μια πραγματιστική θέση. Και το υπογραμμίσατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν ήδη αρκετές υπηρεσίες Ε, όπου εκεί τα θέματα των, της σύγκρουσης των συμφερόντων είναι καθοριστικά. Αν ε, εδώ προσθέσουμε στα πλαίσια αυτού του λογικού φαινομένου και τα τέλη, αν πείτε δηλαδή σε μια υπηρεσία ότι μπορεί να τιμολογεί κάποιες από τις υπηρεσίες της, δεν θα είναι ένδειξη χαρακτήρα από πλευράς της θα αυξήσει σιγά σιγά τις αποδοτικές σε χρήματα αποστολές που τις προσδίδουν οικονομική αυτονομία και θα εγκαταλείψει σταδιακά τις υπηρεσίες τις οποίες δεν είναι αποδοτικές. Κοιτάξτε, η, η υπηρεσία που ασχολείται με τις τράπεζες παίρνει κάποια τέτοια τέλη, εισπράττει τέτοια τέλη. Να σας πω, απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν δώσουμε μεγαλύτερη αυτονομία οικονομική στις υπηρεσίες θα προσανατολιστεί με φυσιολογικό τρόπο προς αυτές. Υπάρχουν βέβαια κάποια τέλη που δεν θα επηρεάσουν τον προσανατολισμό των αποστολών της υπηρεσίας. Θα πρέπει λοιπόν την ιδέα αυτή να την χειριστούμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επιφυλακτικότητα. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή επιτρέπει να προχωρήσουμε λίγο. Και ο τι λέει, παιδί Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ε, χαμογελώ, αλλά δεν ε, γελώ με αυτά που ακούω. Ε, είμαι μάλλον ο πρώτος που έχει επισκεφθεί τις υπηρεσίες. 18 έχω επισκεφθεί ήδη και θα πάω στην 19η σε λίγο. Και πρέπει να πω ότι κάθε τέτοιος οργανισμός είναι τελείως διαφορετικός. Εχθές, ας πούμε, ήμουν στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκα εκεί μία υπηρεσία, το Σεντεφόπ, που ασχολείται με την ε, κατάρτιση, την εκπαίδευση ε, και Νομίζω ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να σκεφτούμε ε, τέτοιου είδους υπηρεσίες να ζητούν τέλη για τις ε, υπηρεσίες που προσφέρουν. Ούτως ή άλλως ε, είναι αναλυτικές οι υπηρεσίες που κάνουν, κάνουν κάποιες δραστηριότητες συντονισμού, ασχολούνται με έγγραφα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση, με την περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση. Ας πούμε, άλλες ε, υπηρεσίες όπως η Europol ή η EASO θα μπορούσαν να ζητούν, να επιβάλλουν τέλη. Υπάρχουν αρκετές ε, υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να ζητούν τέλη για τις υπηρεσίες τους, αλλά δεν το κάνουν. Και νομίζω ότι δεν είναι άσκοπο να μην το κάνουν. Τα καθήκοντα είναι σαφή. Η Άσα είναι μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες της Ευρώπης και βρίσκεται στην κολονία και ελέγχει την ασφάλεια των πτήσεων. Έχουν τόσα πολλά καθήκοντα, τόση πολλή δουλειά που αν είχαν και 100 ανθρώπους ε, παραπάνω στο προσωπικό τους πάλι δεν είχαν πολλή δουλειά να κάνουν. Οπότε κάθε χρόνο ουσιαστικά τους λέμε να μειώσουν το προσωπικό τους. Τέτοιες όμως υπηρεσίες όπως αυτές στην κολονία δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αν δεν έχουν το παραίτητο προσωπικό. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν εδώ η ε, Europol και πέρσι τους είχαμε υποσχεθεί ότι θα, τους, ε, θα έχουν περισσότερες θέσεις ε, εργασίας, περισσότερο προσωπικό. Γιατί η Europol σήμερα δεν δραστηριοποιείται μόνο στην Ευρώπη πρέπει ας πούμε να πάει στην ε, Συρία, πρέπει να πάει στη Λιβύη, πρέπει να πάει στην Τουρκία. Έχουμε αξιωματικούς συνδέσμους στις χώρες αυτές. χρειαζόμαστε και κάποιον στην ε, Χάγη να, για να είναι σε επαφή με όλους τους υπόλοιπους εκτός Ευρώπης. Λέμε ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερα χρήματα ε, στη διάθεση των υπηρεσιών, αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε υποσχέσεις της υπηρεσίας Επίσης, η Eurojust. Γιατί δεν κάνουμε κάτι παρόμοιο με την ε, Eurojust. Η Eurojust είναι πολύ καλή υπηρεσία που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και κλείνω εδώ, Πρόεδρε. Το μέλλον των υπηρεσιών αυτό ποιο θα είναι. Εγώ είπα ότι χτες ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο Σεντεφόπ. Έχουν 91 άτομα προσωπικό. Και πραγματικά είναι αστείο. Κάνουν καλή δουλειά για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, χρειαζόμαστε τις αναλύσεις τους, αλλά δεν είμαστε σε θέση να τους διαθέσουμε το απαραίτητο προσωπικό έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τα καθήκοντα που τους έχουμε αποδώσει. Αυτό είναι το θέμα, γιατί η δουλειά που κάνουν σε αναλυτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, η Europol. Πραγματικά δεν μου αρέσει η κατάσταση. Ε, το 2004 η Τσεχία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, είχαμε πει ότι κάποιες υπηρεσίες που βρίσκονται στα δυτικά της Ένωσης βήμα-βήμα θα έρχονταν προς τα ανατολικά. Τώρα έχουμε δύο υπηρεσίες από το Λονδίνο που πρέπει να μετακομίσουν ίσως θα μπορούσαν να πάνε στην ε, Γερμανία ή στη Γαλλία. Ναι, αλλά η Ρουμανία και η Σλοβακία πόσες υπηρεσίες έχουν. Καμία. Και κλείνω, Πρόεδρε, κλείνω. Όντως, θα πω το τελευταίο. Μιλήσαμε με τους ε, υπευθύνου των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές δημιουργήθηκαν, ναι, και για την ε, εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά πρέπει ίσως να έχουμε ένα κεντρικό όργανο για να τους συντονίσουμε. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εξοικονόμηση χρημάτων. Ευχαριστώ. Θα σας παρακαλέσω όμως να είστε συνοπτικοί γιατί η συζήτηση κάτσε περισσότερο από ό,τι προβλέπαμε. Κύριος Κέλμελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχά, χαίρομαι που όλο και πιο συχνά έχουμε τόσο τεχνικά θέματα στη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα δείγμα αυτό. Εγώ πρέπει να πω ότι ε, έχω μείνει λίγο ενεός. Από τη μία βλέπω ότι έχουμε τα θέματα τα οργανωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Ε, οπότε είτε Χρειαζόμαστε κάποιε υπηρεσίε, κάποιου ε, οργανισμού. πρέπει να δούμε πού είναι καλύτερο να βρίσκονται και πόσο μεγάλοι πρέπει να είναι, τελεία και παύλα. Τώρα, αν θέλουμε να προωθήσουμε τι περιφέρειες, τότε ναι, μπορεί να υπάρχουν καλά ε, επιχειρήματα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την οργάνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να τα αναμειγνύουμε αυτά τα δύο και να τα μπερδεύουμε, νομίζω ότι μα ε, βγάζει από το σκοπό μα. Και έχουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε αυτό το δίλημα. Και γι' αυτό θέλω λίγο να ε, διευρύνουμε το θέμα της συζήτησης. Μονίμως αναρωτιόμαστε αν θέλουμε ε, μια, συνέχεια, μια ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχεται όλο και πιο κοντά. Θέλουμε όλο και περισσότερες ε, ευθύνες, καθήκοντα που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε κατά ανάγκη περισσότερο προσωπικό, που σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα χρειαστούμε περισσότερες υπηρεσίες. Ακριβώς αυτή η συζήτηση δείχνει το πρόβλημα. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου να μπορούμε όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε σε οργανωτικό επίπεδο εναρμονισμένα για όλους και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει καλύτερα ε, σε σχέση με το τι κάνουν επιμέρους τα κράτη-μέλη. Και αυτό υπάρχουν, υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι ακριβώς αυτό το δίλημα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να, να δώσουμε έμφαση. Και υποστηρίζω βεβαίω τον συνάδελφο Γκάιερ και ελπίζω ότι δεν θα πιεστεί πολύ από την πολιτική του ομάδα. Βλέπετε τις συμμαχίες που συσπηρώνει η Ευρώπη. Και τώρα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βρετάνης που έχει καλέσει η κυρία Τομά, τους προσωπικώς, διότι όπως και εγώ, ε, όπως και η κυρία Τομά μάλλον, εκλέγουμε από μια εκλογική περιφέρεια που περιλαμβάνει την Βρετάνη. Καλωσορίζω λοιπόν ε, τους ε, επισκέπτες μας. Ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως προς την ε, γεωγραφική κατανομή των οργανισμών, καταλαβαίνω γιατί ο οργανισμός φαρμάκων πρέπει λόγω χάρη να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα είναι τεράστιο το τίμημα διότι ξέρουμε ότι έχει 800 εργαζομένου ο οργανισμό αυτό στο Λονδίνο και 400 επισκέπτες ανά εργάσιμη ημέρα. Τεράστιο οικονομικό όφελο, οπότε βεβαίω θα υπάρξει χασούρα εφόσον ε, θα χαθεί ο οργανισμός φαρμάκων. Είναι τεράστιο το οικονομικό τίμημα, αλλά εφόσον θέλαμε το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει, είναι... αυτό πρέπει να πληρώσουμε. Ω προ τη χρηματοδότηση των οργανισμών, πρόσφατα στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, εργάνωσα ένα εργαστήριο για το θέμα και κοιτάξαμε τα διάφορα μοντέλα χρηματοδότηση. Ε, του οργανισμού που αυτοχρηματοδοτούνται πλήρω, ε, μερικώ ποιο μέρος πρέπει να αυτό νομίζω ότι σε όλες τι περιπτώσεις είδαμε ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να μπορεί να κάνει για όλους. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι διστάζουν να προωθήσουν την αυτοχρηματοδότηση. Όμως, οι οργανισμοί μπορούν να ε, συγκεντρώσουν ποσά, να κερδίσουν χρήματα και να κάνουν περισσότερα. Μπορούν να δώσουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες πολλέ φορέ. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Υπάρχουν βεβαίω και τα μειονεκτήματα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει διαφάνεια ω προ του εργαζομένου, του εμπειρογνώμονε που απασχολούνται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει πλεόνασμα και τι γίνεται με αυτό. Το πλεόνασμα που πηγαίνει είναι ένα θέμα που πρέπει να το βλέπουμε αλλά μέσα σε όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει να αποκλείσουμε κανένα μοντέλο χρηματοδότηση. Θα πρέπει να δούμε τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά και να είμαστε βέβαιοι ότι χρηματοδοτείται όπω πρέπει, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για του πολίτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βόν. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει την δική της άποψη σε αυτή την προκεχωρημένη ώρα της πρωίας. Διότι έχω την εντύπωση Είμαι κλεισμένο μένα, αλλά για τρίτη φορά συμμετέχω σε συνεδρίαση για του οργανισμού. Έχω την εντύπωση ότι λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταφέρει να, λάβει τις σωστές, να λαμβάνει τι σωστέ αποφάσει. Πώ γίνεται. Πώ γίνεται να μην λαμβάνονται αποφάσει. Υπάρχει θέμα συνέπεια, υπάρχει θέμα τη λειτουργία. Θέλετε να μα ε, ενημερώσετε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας δώσω κάποιους αριθμούς στην αρχή, τους οποίους θα βρείτε κιόλας στην πρόταση προϋπολογισμού για το 18. Θα συμφωνήσω καταρχάς με αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι το 18 είναι η τελευταία χρονιά για τη μείωση του προσωπικού. Η πρόταση που κάνει η Επιτροπή για τον προϋπολογισμό του 18 ολοκληρώνει το μείον 5% για όλες συνδυαστικά τις υπηρεσίες εξωτερικές. Η Επιτροπή είπε ότι τερματίζουμε εδώ και δεν θα συνεχίσουμε με περαιτέρω μειώσεις πέραν του 18. Τώρα, πώς αυτές οι μειώσεις του προσωπικού επιτυγχάνονται. Υποτίθεται ότι έπρεπε να μειώσουμε κατά 254 πρόσωπα το προσωπικό των υπηρεσιών μέσα σε 5 χρόνια. Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει 700 ε, τόσες θέσεις παραπάνω από τον στόχο αυτό. Αντί λοιπόν να μειώσουμε κατά 5% είμαστε σε αύξηση 7,5%. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, ε, έχουμε το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης. Τα τελευταία πέντε χρόνια αυξήσαμε, προτείναμε και έγινε δεκτό, να αυξήσουμε 520, με 522 θέσεις το Frontex, 273, η Άσο 157 και άλλες 6 υπηρεσίες. Για θέματα ασφαλείας, η αρχή επί του προϋπολογισμού μετά από πρότασή μας δέχτηκε 91 επιπλέον θέσεις πέραν των προβλεπομένων του στόχου μείωσης. Αποκλειστικά για τη Europol, σχεδόν αποκλειστικά. Και τρίτον έχουμε το πιλωτικό για τον ΕΑΣΑ, όπου ελέγχουμε σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να εξαρτηθεί ο αριθμός του προσωπικού από την εξέλιξη του, ε, της εργασίας, των δράσεων και των αποστολών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής και στα πλαίσια της πρότασης του 18 είναι για την ΕΑΣΑ αύξηση 36 υπαλλήλων. Τελικό συστατικό αυτής της απόκλησης, αν θέλετε, στους στόχους είναι τα λεγόμενα top-ups, τα οποία συμφωνήθηκαν τα τελευταία χρόνια για 10 υπηρεσίες και τα οποία τα τελευταία 4 χρόνια, δεν έχει υπάρξει συνδιαλλαγή για το 18, 56 θέσεις υπαλλήλων με τα top apps. Οι εκπρόσωποι λοιπόν, ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών αναφέρθηκε σε αυτά και είναι αλήθεια ότι ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές έχουν μειώσει το προσωπικό τους με πάνω από 5%. Είναι 12 αυτές οι υπηρεσίες που μειώσαν 10% το προσωπικό τους Συμπληρωματικά υπήρξαν δύο επιπλέον υπηρεσίες οι οποίες πέτυχαν μία μείωση όχι 10% δεν ήταν στόχος αυτό το 5% από τις 32 λοιπόν υπηρεσίες υπάρχουν 14 οι οποίες πέτυχαν την μείωση του 5%. Όλες οι άλλες για πολύ συγκεκριμένους λόγους τους οποίους συμφωνούμε ε, είτε αυξήθηκαν είτε ε, μειώθηκαν κατά 5%. Τώρα για τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται και αποτέλει. Είναι 8 οι υπηρεσίες αυτές οι οποίες είτε χρηματοδοτούνται επιμέρους, η ΕΚΑ, η ΆΖΑ και τα φάρμακα. Μερικά λοιπόν αυτοχρηματοδοτούνται. Υπάρχουν ε, δύο επίσης οι οποίες χρηματοδοτούνται πλήρως, Αλικάντε και η Υπηρεσία για τα, την Ευρεσιτεχνία. Υπάρχουν επίσης και άλλες οι οποίες χρηματοδοτούνται κατά 60% από εθνικές συνεισφορές και κατά 40% από τον προϋπολογισμό της κοινότητας. Στόχος είναι η αντικατάσταση των εθνικών συμμετοχών στο μέλλον από συμμετοχές της ε, βιομηχανίας, ε, της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα. Τώρα, να αυξήσουμε την δυνατότητα των υπηρεσιών να εισπράττουν τέλη είναι μια δυνατότητα η οποία μπορεί να εξεταστεί και ήδη εξετάζεται και στα πλαίσια της θεσμικής ομάδας, της διοργανικής μάλλον ομάδας. Άκουσα τον κύριο Γκάγερ να είναι θετικός. Φυσικά έχουμε την ευθύνη εμείς για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να, να ελέγξουμε, να συμπιέσουμε τις διοικητικές δαπάνες και να παρακολουθήσουμε από πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις των τελών αυτών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι υπερβολές. Αλλά μέχρι τώρα το σύστημα φαίνεται ότι λειτουργεί σχετικά ικανοποιητικά. Τελειώνοντας, να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για την έδρα των επιχειρήσεων. Τα μέλη της Επιτροπής σας έχουν εκφράσει επανειλημμένα τις απόψεις τους για κάποια προβλήματα και κάποιες δυσκολίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το θέμα αυτό να συζητηθεί στα πλαίσια των συστάσεων τις οποίες θα καταθέσει η Διοργανική Ομάδα Εργασίας στις επόμενες συναντήσεις της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει ε, με συγκεκριμένες ιδέες προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρόταση σύμπτυξη ΣΥΠΟΛ και Europol δεν έγινε δεκτή ούτε από το Συμβούλιο ούτε από το Κοινοβούλιο. Και επίσης οι δύο έδρες της ΝΙΣΑ να συμπτυχθούν σε μία είναι κάτι το οποίο θα επανεξεταστεί όταν κάνουμε εμείς ε, την πρόταση για την αναθεώρηση της ΕΝΙΣΑ ε, στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, ε, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις εξηγήσεις, οπότε η κατάσταση θα αλλάξει και θα μετατραπεί. Κύριε Ντεπρέ, πολύ γρήγορα. Ε, ναι, δεν θέλω να ξανανοίξω τη συζήτηση. Θέλω απλώ να συνεισφέρω στα προηγούμενα. Ραντεβού τότε σε μια επόμενη συνεδρίαση για τους οργανισμούς. Κύριε Σιγητά, Υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν και να μετατραπούν. Το Συμβούλιο μπλοκάρει τα περισσότερα όμως. Εδώ δεν μιλάμε για οργανισμό σε αυτή την περίπτωση, αλλά για θέση δικαστού. Επί τέσσερα χρόνια το Συμβούλιο δεν συμφωνούσε για να ε, καλυφθεί μια θέση και τελικά πρόβλεψε 28. Γιατί, Γιατί υπάρχουν 28 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε ενδεχομένω, κύριε Σιγητά, να επικοινωνούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μα, διότι μόνο κοινή γνώμη μπορεί να πιέσει το Συμβούλιο να δράσει. Για κάποιε μη κανονικότητε. Για κάποιε δυσλειτουργίε πρέπει να φροντίσουμε να προφέρονται στα μέσα μαζική ενημέρωση για να ασκηθεί πίεση και να λαμβάνονται αποφάσει. Κύριε Ισηγητά, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα να πω εγώ μόνο. Ούτε οι υπηρεσίε, ούτε εγώ να έχουμε την ιδέα ότι, κάποια, ότι κάθε υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τέλη. Ο συνάδελφος έδωσε κάποια ε, παραδείγματα υπηρεσιών που, θα μπορούσαν, ε, που δεν θα μπορούσε μάλλον αυτό να λειτουργήσει καθόλου. Υπάρχουν λοιπόν ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων καταστάσεις όπου πολλές υπηρεσίες που έχουν, παρέχουν υπηρεσίες στα θεσμικά όργανα δεν είναι σε θέση για διάφορους λόγους να επιβάλλουν τέλη. Όταν όμως επιβάλλουν, ε, εγώ μίλησα για ε, υπηρεσίε ε, σε τρίτου. και εκεί μιλούμε για τη βιομηχανία κυρίω αυτό, μπορούμε να το εξετάσουμε. Αν δούμε ότι ας πούμε μπορούμε να, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη επίδεξη των στόχων της Επιτροπής. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι το θέμα της κατανομής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η πιθανή αντίφαση των δύο επιχειρημάτων. Την αρχή της δίκης κατανομής των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στα κράτη-μέλη. Αυτό βεβαίω είναι σημαντικό και το σέβομαι. Απ' την άλλη, έχουμε τη συζήτηση που γίνεται συνέχεια για την απόδοση, την συγχώνευση, τη συνέργεια, τη συνεργασία. Και νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση δεν μπορούμε να την κάνουμε με τέτοιο τρόπο που τα επιχειρήματα να προκύπτουν ανάλογα από το ποια αρχή πλήττεται. Ο Χωσέ Μανουέλ και εγώ ε, συνήθως είμαστε μια καρδιά και μια ψυχή. Ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, συγκέντρωσης όλων στις Βρυξέλλες, αλλά αν πούμε ότι θέλουμε την ε, κατανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το Κοινοβούλιο και αυτή εδώ η Επιτροπή είναι αυτή που θα πρέπει να κρατηθεί και τα θέματα κατανομής των υπηρεσιών και των ευρών να, για να λάβει τις δύσκολες ίσως αποφάσεις που θα χρειαστούν. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι κάποιος εδώ στην υπηρεσία, που, στην αίθουσα που να λέει ότι κάποιος από την ε, ΕΜΠΑ ή την EMA από το Λονδίνο θα πρέπει οπωσδήποτε να πάνε είτε στη Σλοβακία είτε στη Ρουμανία. Νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλες προσφορές εδρών. Ας πούμε την ΕΜΠΑ θα μπορούσαμε να την έχουμε μαζί με μια ε, υπηρεσία ελέγχου, οικονομικού ελέγχου. Ναι, γιατί όχι. Το λέει και η Κλαούντια, γιατί όχι. Αυτό ακριβώς όμως συζητούμε. Ποια είναι η αρχή που θα πρέπει να υπηρεσχύσει. Υπεραμεινόμεθα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ναι, άρα υπάρχουν πολλοί που θα το πράξουν αυτό και εγώ θα το κάνω αυτό. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει δύο υπηρεσίες. Υπάρχουν άλλα που Επίσης έχουν πέντε υπηρεσίες στην επικρατεία τους και ζητάνε και έκτη, χωρίς πρόβλημα και κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί η, τελική απόφαση. Ποιος αποφασίζει, πού θα πάει η, η υπηρεσία, γιατί να πάει στο Βουκουρέστι ας πούμε ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Αυτά λοιπόν είναι θέματα σημαντικά και είναι λίγο κουραστικό όταν η έδρα μιας υπηρεσίας και ο συνάδελφος από την Κομισιόν το είπε, αυτή εδώ η Επιτροπή ήταν που αποφάσισε το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, όχι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, συγγνώμη, η ε, υπηρεσία για την αστυνομία να πάει στην Χάγη και να ενισχυθούν οι συνέργειες. Η Ολομέλεια έχει αποφασίσει διαφορετικά, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει διαφορετικά, η υπηρεσία πήγε στην Βουδαπέστη. Ε, ναι, ναι, κάναμε σωστά την κατανομή, αλλά δαπανίσαμε έξτρα χρήματα. Και πρέπει να πω ότι μονίμως η μία ε, αρχή μπορεί να αντιπαρατεθεί με την άλλη. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε η Επιτροπή Προπολογισμών. Και καθήκον μας είναι να παρακολουθούμε κατά πόσον ο κάθε οργανισμός ανταποκρίνεται στην ε, απέτηση τη θέμενης αξίας. Καταλαβαίνουμε ότι περίπου κάθε χώρα θα έπρεπε να έχει έναν οργανισμό, αλλά εδώ είμαστε για να βεβαιωθούμε ότι οι δημόσιες δαπάνες, κάθε ευρώ που δαπανούμε, κάθε ευρώ που ζητούμε από τον φορολογούμενο, αμέσως ή εμέσως ε, μέσω των εθνικών κρατών, ε, εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον. Ο κύριος ο οποίος εκπροσώπησε τους οργανισμούς, ε, σήμερα το πρωί θέλει να πει λίγα λόγια. Θέλετε να μας πείτε τι μαθήματα αντλείτε, τι διδάγματα από την σημερινή ανταλλαγή και συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εάν μου επιτρέπετε, πολλά πολιτικά ζητήματα συζητήθηκαν εδώ και εμείς ως οργανισμοί δεν μπορούμε να ε, επηρεάσουμε αυτές τις συζητήσεις πόσες, ε, πόσους πόρους θέλετε λόγω χάρη να αφοσιώσετε στην ΕΦΣΑ, την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα απαιτούν και πόρους για να εκτελεστούν. Αν δεν έχουμε πόρους, δεν θα μπορούμε να φέρουμε σπέρα στις αποχρεώσεις μας. Ω προ τι έδρε τη συγχωνεύσει οργανισμών, όπω είπατε, είναι πολιτικό το ζήτημα, κατεξοχήν. Αυτό που εμεί μπορούμε να κάνουμε και αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε τι κοινέ υπηρεσίε να τι προωθούμε, ώστε να εξισορροπήσουμε, εάν μπορώ να το πω έτσι, το μειονέκτημα της γεωγραφικής, ε, του γεωγραφικού κατακαιρματισμού στην Ευρώπη το ότι βρισκόμαστε σε πολλά διαφορετικά σημεία, ε, Υπηρεσίε σε ανθρώπινους πόρους, σε προσλήψεις, σε επικοινωνία και πληροφορική, σε ανακούφιση από φυσικέ καταστροφές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι και το καθήκον μας. Και γι' αυτό έχουμε διοριστεί ω ε, διευθυντέ και εκτελεστικοί διευθυντέ των οργανισμών. Και κάτι ακόμη που θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί είναι η διακυβέρνηση, η σωστή διαχείριση των οργανισμών. Εκεί δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε το Συμβούλιο. Εκεί πρέπει να δούμε πώ θα προσφέρουμε ευελιξία στην διαχείριση των οργανισμών και να χρησιμοποιούν του πόρου του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν μου επιτρέπετε, θα πω ότι ο άριστο τρόπο δεν είναι να μετράμε τα κεφάλια των εξωτερικών συνεργατών ή των συμβασιούχων, και να βάζουμε ε, όριο στον αριθμό συμβασιούχων που μπορεί να απασχολήσει ένας οργανισμός. Το ερώτημα είναι πώς θα έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελο σε σχέση με το κόστος των οργανισμών. Πρέπει δηλαδή να βασιζόμαστε σε μια προσέγγιση ε, σχετική με τις επιδόσεις, με το όφελος παράγεται για να μπορεί και η διεύθυνση του οργανισμού να κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι η δουλειά των μάνατζερ, γι' αυτό μας διορίζουν και μας εκλέγουν για πέντε χρόνια. Θέλουμε να φέρουμε εις πέρας ένα έργο, να κάνουμε τη δουλειά μας ε, με ευσυνείδητο τρόπο. Εάν δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας για πέντε χρόνια, θα μας πετάξετε έξω και θα χάσουμε τη δουλειά μας. Γι' αυτό αφήστε τους μάνατζερ να κάνουν τη δουλειά τους, να μπορούμε εμείς να μετράμε την αξία μας, το τι παράγουμε σε σχέση με αυτά που λαμβάνουμε. Θα καλύπταμε πολλές ανεπάρκειες, αν μας επιτρέπατε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να είμαστε μαζί σας σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα της διακυβέρνησης των υπηρεσιών είναι βασικό και για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο έχετε περιθώρια αύξησης του επίπεδου ελευθερίας επιλογής στόχων της κάθε υπηρεσίας. Νομίζω, νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έχετε περισσότερες ευθύνες, περισσότερη ελευθερία και να υπάρχει αυθεντική προστιθέμενη αξία. Αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε την επόμενη φορά τις θετικές εξελίξεις. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των υπηρεσιών. Ευχαριστώ λοιπόν τους εκπροσώπους για την παρουσία τους. Ο κύριος Ντεπρέ, θέλετε να μας μιλήσετε για το αίτιας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να εξηγήσω καταρχάς τι είναι το αίτιας. είναι ένα νέο σύστημα ενημέρωσης σε μεγάλη κλίμακα που έχει σαν στόχο τη διαχείριση της εκ των προτέρων αδειοδότησης για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που εξαιρούνται από το σύστημα των θεωρήσεων. Όλοι αυτοί οι πολίτες θα πρέπει να καταθέσουν ε, μια αίτηση εκ των προτέρων για να γνωρίζουν αν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύστημα σαν αυτό το ΕΣΤΑ των Ηνωμένων Πολιτειών και αντίστοιχα στον Καναδά και την Αυστραλία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να έλθουν στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αεροπλάνο, με πλοίο, με τρένο, με αυτοκίνητο θα πρέπει να ζητήσουν εκ των προτέρων την άδεια. Αυτό ακούγεται λίγο σαν κάτι να φοβίζει, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ε, θα υπάρξει μια βασική αρχή την οποία θα διαμορφώσει σε τεχνικό επίπεδο η ΕΝΙΖΑ και θα διαχειριστεί τον Φορτεξ. Ε, ε, σε αυτή την περίπτωση που κάποιος καταθέτει, αν θέλετε, το ερώτημα σε ένα μεγάλο ποσοστό θα παίρνει την απάντηση κατά 95% σε 5 δευτερόλεπτα. Το 5% θα γίνεται αντικείμενο ανάλωσης αν υπάρχουν προβλήματα ομονιμίας σαν παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια εντοπισμού των προσώπων αυτών. Και επίσης όλα αυτά θα ελέγχονται από τις εθνικές μονάδες. Κάθε χώρα θα έχει τη δική της εθνική μονάδα που θα διαχειρίζεται τις προβληματικές αιτήσει, είτε γιατί θα είναι η χώρα εισόδου, είτε για άλλους λόγους τα θέματα αυτά δεν έχουν ακόμα όμως καθοριστεί πλήρως στο Συμβούλιο. Συνολικότερα λοιπόν θα έλεγα ότι το 95% των περιπτώσεων δεν είναι προβληματικά και 5% θα αντιμετωπίζονται ατομικά όχι από πληροφορικά συστήματα, αλλά από συγκεκριμένους υπευθύνους υπαλλήλου έτσι ώστε να έχουμε τις πληροφορίες τις οποίες θέλουμε. Εμείς είμαστε η Επιτροπή Προϋπολογισμών, το σύστημα αυτό έχει ένα κόστος, η εφαρμογή του συστήματος ε, υπολογίζεται σε 212 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνουμε το κόστος λειτουργίας και ανάπτυξης ε, του κεντρικής μονάδας ε, και της ενσωμάτωσης των υπαρχουσών εθνικών υπηρεσιών. 212 εκατομμύρια. Μετά το κόστος θα είναι 85 εκατομμύρια το χρόνο αλλά εδώ θα έχουμε με τα τέλη και τις συνδρομές να τα καλύψουμε αυτά. Δεν θα κοστίσει κάτι και θα βελτιώσω την κατάσταση έτσι ώστε να διασφαλίσω επιπλέον έσοδα. Το σύστημα λοιπόν αυτή στιγμή σε κινήσει θα είναι αυτόνομο οικονομικά. Ταυτόχρονα γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση και μια μικρή αντιπαράθεση ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και ε, ε, εμάς αν θα πρέπει να δώσουμε εξωτερικά δικαιώματα ής τελών ε, χωρίς να υπάρξει ξεκάθαρη νομική πράξη. Εδώ υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Τώρα για το δημοσιονομικό κομμάτι, εγώ αυτό το οποίο προτείνω είναι το εξή. Τα κράτη-μέλη θα τους κοστίσει κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος. Είναι πως εγώ λέγω ότι το κόστος λειτουργίας των εθνικών μονάδων να λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας. Αυτό θα α, ε, διευκολύνει κάπως το χρέος, τα χρέη μάλλον των κρατών μελών. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάθε αίτημα εκ των προτέρων αδειοδότησης που κανονικά θα πρέπει να ισχύσει η πενταετία, δηλαδή κάθε πέντε χρόνια πρέπει να ζητάει κανείς την άδεια, θα κοστίζει 5 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι η διάρκεια δεν είναι το πρόβλημά μου βέβαια ουσίας, αλλά η διάρκεια αυτής της αδειοδότησης να είναι 3 και όχι 5 χρόνια. Γιατί λόγω των προβλημάτων τα οποία γνωρίζουμε σήμερα, στα προβλήματα ασφαλείας εννοώ, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται τάχιστα. Ω εκ τούτου λοιπόν η διάρκεια τη πενταετία, η πενταετή συγγνώμη διάρκεια δεν είναι κατάλληλη και πρέπει νωρίτερα να επανελέγχεται. Επίσης θεωρώ ότι το κόστος αδειοδότησης θα πρέπει να είναι 10 ευρώ. Θα σας εξηγήσω γιατί προτείνω 10 και όχι 5. Αν δείτε το σύστημα σε άλλες χώρες τι βλέπετε. Στις ΗΠΑ Μία εκ των προτέρων αδειοδότηση κοστίζει 14 ευρώ για δύο χρόνια, 7 ευρώ το χρόνο. Η Αυστραλία είναι 16 ευρώ τον χρόνο. Και αν δεχθείτε την πρότασή μου που είναι 10 ευρώ ε, για 3 χρόνια είναι 3,33 ευρώ κατέτος κόστος τι μπορεί να δώσει το σύστημα αυτό εφόσον γίνει δεκτός ο μηχανισμός τον οποίο προτείνω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 39 εκατομμύρια πολίτες τον χρόνο που έρχονται, είναι υπολογισμός της Επιτροπής, τότε πολλαπλασιάζεται ε, το ποσό με το 10 και καταλαβαίνετε ποιο είναι το ποσό το οποίο μπορούμε να εισπράξουμε. Προτείνω επίσης ότι κάθε επιπλέον πόρος, ο οποίος θα παραμείνει διαθέσιμος μετά από την κατανομή κάλυψης ε, των δαπανών, θα πρέπει να αποδίδεται στην κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Και μιας και αυξάνω ουσιαστικά το κόστος, προτείνω αντισταθμιστικά ορισμένες κατηγορίες να την χάνουν εξαιρέσεων Ζητώ σαν παράδειγμα οι καθηγητές, διδάσκοντες και φοιτητές ε, στη ζώνη Σέγγεν να εξαιρούνται. Το ίδιο και για τους ερευνητές και το ίδιο και για τους εκπροσώπους των ΜΚΙΟ. Προτείνω επίσης να ευθυγραμμιστεί η εξαίρεση κόστους για τα παιδιά μέχρι τα 12 όπως ακριβώς προβλέπεται αν θυμάμαι και για το σύστημα των θεωρήσεων το σημερινό. Οπότε γιατί να έχουμε διαφορετικό σύστημα για αυτούς που α, υπόκεινται στο σύστημα των θεωρήσεων και για αυτούς που απαλλάσσονται. Λοιπόν, συμπερασματικά πρόεδρε, είμαι υπέρ του συστήματος αυτού, αν και δεν είμαστε υπεύθυνοι από της ουσίας. Δεύτερον, σας εξήγησα πώς λειτουργεί. Τρία, σας εξήγησα πόσο θα κοστίσει. Και τέσσερα, σας εξήγησα ποιες είναι οι τροπολογήσεις τις οποίες προτείνω προς όφελος των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Όλα αυτά ήταν ε, απολύτως σαφή. Και τώρα να ζητήσω... Ε, πρόεδρε, με συγχωρείτε μια ερώτηση. Δεν άκουσα Πόσο έποτε θα κοστίσει στον προπολογισμό τη Ένωση 212 η επένδυση και 85 ε, το κόστο λειτουργία Το χρόνο. Ετησίω, ετησίω. Και πολλά εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Εάν ζητήσουμε 30 εκατομμύρια το χρόνο και παίρνουμε 10, ε, πρέπει να κάνετε τον πολλαπλασιασμό. Με συγχωρείτε, 90 είναι το αποτέλεσμα, όχι 90 στα βέλγικα, είμαι επαρχιώτης. Ε, ε, μπορείτε να προσθέσετε και τους μαθητευόμενους εδώ, τους ασκούμενους. Ο κύριος Σαρβαμά, ο οποίος είναι σχεδόν εισηγητής για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Ντεπρέ. Ειλικρινώς τον ευχαριστώ για την ε, έκθεση. Ζεράρ, με τα χαράς να σου πω ότι στα βασικά σημεία συμφωνώ με όσα είπες. Απλώ να προσθέσω το εξή. Διερωτώ με γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι τόσο μετριοπαθή ε, στο ποσό. Βλέπουμε όλοι με έναν απλό υπολογισμό ότι αυτό δεν είναι και μια μηχανή που θα παράγει χρήμα ούτω ή άλλω. Αλλά το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να καλύψουμε το κόστος. Εάν δούμε τι κάνουν άλλες χώρες σχετικά, νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο να είναι το ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ. Επίσης με ένα τριετή κύκλο. Κάποια στιγμή σαφώ θα υπάρξει επιβράδυνση, επιβράδυνση και όπως σωστά είπε ο Πρόεδρος, είναι δύσκολο να πούμε πόσα χρήματα, τι ποσό θα μας έρχεται ως κέρδος. Πάντως δεν θα είναι τίποτα τεράστια τα ποσά ούτως ή άλλως, αυτό είναι σαφές. Ω προ τι αλλαγέ λοιπόν αυτές νομίζω είναι σημαντικό να γίνουν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης εκτιμώ τι τροπολογίε σας Πρέπει να αποστείλουμε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τους φοιτητέ, ερευνητέ, διδάσκοντες όμως έχω και μια-δυο οι εγκρίσει για ταξίδια, μετακινήσει για αυτού του ανθρώπου, για αυτήν την ομάδα ανθρώπων, θα ισχύει για ένα μόνο ταξίδι ή για όλη την τριετία. Διότι ω προ την ασφάλεια δημιουργείται με ένα παραθυράκι εδώ. Για παράδειγμα, όταν οι φοιτητέ ή οι εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικού οργανισμού, εάν επί τρία χρόνια μπορούν να ταξιδεύουν δωρεάν, ξέρετε τι γίνεται με του εργαζομένου τη μη κυβερνητικέ οργανώσει. Αλλάζουν δουλειά συνέχεια. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ε, να είναι κάτι που ελέγχεται και να είναι και καλό το σύστημα, όπως το προτείνει η εκθεσή σας. Λέτε στην έκθεση η ε, μορφή οργάνωση πρέπει να αλλάξει. Να φανεί λοιπόν ότι εντάξει θα λάβουμε μέρημνα για αυτές τις κατηγορίες, αλλά ταυτόχρονα θα προσέχουμε πώς θα λάβουμε αυτή τη μέρημνα και πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σε σχέση με την ε, ε, διατήρηση του συστήματος αίτιας. Νομίζω ο δικός μας σκοπός είναι να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του αίτιας, του συστήματος αυτού. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός, θεωρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της ίδιας άποψης. Θα ήθελα να σας πω ότι σημειώνω τις προτάσεις για αλλαγές στο σχέδιο γνωμοδοτησής και νομίζω ότι η σημαντικότερη αλλαγή που χρειάζεται είναι ο τρόπος που θα αξιοποιούνται τα έσοδα αυτού του συστήματος και η χρήση των υπολοιπόμενων ε, ποσών αφού έχουν καλυφθεί όλα τα κόστη λειτουργίας. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές που θα έπρεπε να τις προσέξουμε πιστεύω και με τροπολογίες θα κοιτάξουμε να τις θίξουμε. Δηλαδή, πρώτον να δούμε τις κατηγορίες των ε, ανθρώπων που θα λαμβάνουν αυτή την έγκριση, αυτή την εξουσιοδότηση. Πρέπει να ορίσουμε και ένα όριο ηλικία. Και έπειτα, ε, οπωσδήποτε, πρέπει να συζητήσουμε για το ποσό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 ευρώ, εσείς 10, πρέπει να βρούμε ένα ε, μια λύση που να είναι η καλύτερη δυνατή και για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και για τους υπηκόστριτων τρίτων χωρών που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ισχύει και για τη διάρκεια ζωή τη άδεια άδειας, της αλλά να πω εδώ εν παρενθέσει ότι η αναθεώρηση του κεκτημένου Σέγγεν και η ενδεχόμενη απλούστευσή του είναι καλοδεχούμενη, ιδίως στο πλαίσιο όπου η Ρουμανία και η Βουλγαρία κάποια στιγμή θα πληρούν τα κριτήρια για να συμμετέχουν στο Σέγγεν. Ε, αυτό το έχω πει επανειλημμένο στην Επιτροπή Προπολογισμών. Χρειαζόμαστε ένα Σέγγεν ισχυρό. Ένα χώρο Σέγγεν ισχυρό που να συγκεντρώνει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό του. Έτσι το σύστημα αίτια θα λειτουργεί ιδανικά. Ω συμπρόεδρο τη ομάδα μου για την ε, πρόθεση του ευρωπαϊκού τουρισμού εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι έμεσε και άμεσε συνέπειε που θα έχει η πρόταση αυτή, η πρόταση του κανονισμού για τον τουρισμό. Θέλουμε να προσελκύσουμε τουρίστε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, στο ποσό που θα προβλέψουμε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και διαδικασία screening για λόγους προφύλαξης. Να είμαστε βέβαιοι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ό,τι τίμημα ζητούμε από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ανάλογο με τον σκοπό του ταξιδιού και να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε με το απόρριτο και την εμπιστευτικότητα ούτε με την προστασία των δεδομένων. Επίσης, οι τουρίστες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχουν μια θετική εμπειρία. Αυτό θέλουμε να αποκομίζουν. Και είναι σημαντικό για να, ε, και να, να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι ταξιδεύουν για διαφορετικούς λόγους, για σπουδές, για δουλειές, ε, για τουρισμό, αλλά θέλουμε η Ευρώπη να βρίσκεται στι πρώτε θέσει του παγκόσμιου τουρισμού, διότι υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό με τον υπόλοιπο κόσμο, την Ασία, την ε, Κεντρική Αμερική και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να πληγεί αυτός ο κλάδος της οικονομίας εάν δεν λάβουμε συνετές αποφάσει. Επίση να πω τα εξή η προθεσμία για την απόκτηση τη εξουσιοδότηση τη έγκρισης, ε, εάν ο κατάλογος των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι πολύ μακροσκελής. Αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόφαση των τουριστών να έρθουν ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φρονώ ότι είναι σημαντικό κάτι που δεν φάνηκε ανάγλυφα από τη συζήτηση που είχαμε εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών ακόμα, ότι όλη αυτή η υπεράσπιση και η ομιλία υπεράσπισης του τουρισμού και του ευρωπαϊκού τουρισμού είναι πολύ σημαντική γιατί ε, ο τουρισμός είναι 5% του ευρωπαϊκού ΕΠ και έχει να καλύψει 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν ε, που σας επισημαίνω εδώ στη συζήτηση θα συμπεριλαμβάνονται στι τροπολογίε των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ελπίζω ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έγκριση του κανονισμού αίτιας. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλους σκιώδει εισηγητέ εδώ στην αίθουσα. Προσκαλώ λοιπόν τους ε, συναδέλφους να λάβουν το λόγο αφού τα επιθυμούν. Εφόσον όχι, ας μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντεπρέ για την στήριξή του προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως πρώτα να διευκρινίσω... Ναι, μόνο μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Πόσο κοστίζει η ανάκτηση αυτού του τέλους, το 5 και 10 ευρώ. Υπάρχει διοικητικό, διοικητική διαδικασία για την ανάκτηση. Κανονικά πληρώνεται με πιστοτική κάρτα. Δεν υπάρχει κόστος, συγκεκριμένο κόστος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το κόστος του συστήματος, όπως εξηγήθηκε από τον κύριο Ντεπρέ, θα είναι 85 εκατομμύρια ετησίως. Για να είμαστε απολύτως σαφείς ακόμη και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εισόδημα που θα παράγει το ΕΤΙΑΣ θα είναι υπεραρκετό για να καλύπτει το κόστος λειτουργίας του. Μιλάμε για 39 εκατομμύρια ετήσεις ετησίως 5 ευρώ αναέτηση, οπότε περίπου 200 εκατομμύρια εισόδημα ετησίω για να καλύψουμε το εκτιμόμενο κόστος λειτουργίας 85 εκατομμυρίων. Δηλαδή υπερδιπλάσιο το εισόδημα. Ε, σημειώνουμε τις προτάσεις του κυρίου Ντεπρέ βεβαίω, να διπλασιάσουμε κι εμείς το εισόδημα που προβλέπεται να αποκομιστεί. Αυτό προφανώς θα συζητηθεί στους τριμερείς διαλόγους σε κατοπινή φάση. Το κατά πόσον είναι καλή ιδέα να προχωρήσουμε με την εξαίρεση από το τέλος αυτό, ίσως να είναι αναγκαίο. Εάν ληφθεί η απόφαση να αυξηθεί μάλιστα το κόστος καθέτησης, άποψη όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι στη δική μας την πρόταση ένα κόστος 5 ευρώ αναέτηση για 5 χρόνια δεν θα είναι απαγορευτικό και δεν υπάρχει και λόγος να εξαιρεθεί ή από την καταβολή αυτού του τέλους. Σημειώνουμε την πρόταση του εισηγητή να διευρύνουμε το πεδίο για το εξωτερικό ε, εισόδημα για ειδικό σκοπό και ευχαριστούμε τον κύριο Ντεπρέ που στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, να ε, συμφωνεί με την πρόταση για εξωτερικό ε, εισόδημα για ειδικό σκοπό, κάτι το οποίο δεν εγκρίνεται για την ώρα από το Συμβούλιο. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την ιδέα διεύρυνσης του πεδίου, κάτι που σίγουρα θα συζητηθεί περαιτέρω. Πιστεύω ότι ολοκλήρωσα τα σχολεία μου με αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεπρέ, έχετε την τελευταία κουβέντα να μας την πείτε. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο να διευκρινίσω, κυρία Ταπαρντέλ, και σε ένα βαθμό, κύριε Σαρβάμα, ότι περιορίστηκα στις δημοσιονομικές πτυχές. Εσείς καλύψατε πάρα πολλά άλλα στοιχεία με τα οποία συμφωνώ και επειδή είμαι εισηγητής και ομοδότηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα κάνω εκεί τις σχετικές προτάσεις και τροπολογίες. Σας ευχαριστώ κύριε Σαρβαμά. Εάν καλά κατάλαβα, 10 ευρώ για τρία χρόνια είναι κάτι που θα σας άρεσε. Επίσης θέσατε μια ερώτηση για την διάρκεια της εξαίρεσης. Όντω είναι ένα σημείο ε, το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχω σκεφτεί. Θα κοιτάξω να το σκεφτώ και να σα απαντήσω. Ναι, γιατί ένα φοιτητή δεν είναι αναγκαστικά φοιτητή τρία χρόνια. Ναι, αλλά όταν έχει πάρει κανεί έγκριση για ταξίδι σε 27 ε, κράτη ε, και είναι 18, το να έχει την ίδια έγκριση στα 21 το δεν αλλάζει και πολλά. Τέλο πάντων, είναι πολλά αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ταπαρντέλη περιμένω διακαώ τι τροπολογίε, ιδίω σε σχέση με το που αναφέρατε για την αναλογικότητα, αλλά μην τα υποβάλλετε εδώ, διότι εδώ είμαστε αρμόδιοι για τα θέματα τα δημοσιονομικά, του προπολογισμού. Οπότε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Πρόεδρε, θα περιμένω τι προτάσει, τι τροπολογίε των διαφορών συναδέλφων. Σα ευχαριστώ. Διευκρινίζω ότι οι τροπολογίε θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο 19 Ιουλίου στι 12 το μεσημέρι. Ε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών προβλέπεται 30 και 31 Αυγούστου και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, καθήλυνα αρμόδια, θα ε, εγκρίνει την δική της έκθεση ε, και θέση τον Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλες και όλους σας. Ευχαριστώ τον συγκεκριτή μας, τον κύριο Ντεπρέ. Και τώρα, καλώ τον κύριο Σαρβαμά Όχι, ο κύριος Μάνκα είναι. Κύριε Μάνκα, έλεγχος. Μα ναι, είμαστε στη σωστή σειρά. Είπατε το επόμενο. Α, ναι, όμως ο κύριος Μάνκα έχει μια ε, ηλυμένη υποχρέωση. Εάν θέλετε κύριε Σαρβαμά, να του δώσουμε την προτεραιότητα. Έλεγχος δαπανών και παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων των εγγύσουν για την νεολαία. Κύριε Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σάβαμα που μου δίνει το λόγο να κάνω πρώτο στην παρέμβασή μου. Ο στόχο των εγγύσεων για την νεολαία είναι βεβαίω η υψηλή ποιότητα εργασία για όλους τους ε, νέου. η καλύτερη κατάρτιση, μετεκπαίδευση, μια θέση ε, μαθητείας ε, εντός τεσσάρων μηνών. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει από την από τους διάβλους επίσημης εκπαίδευσης ή βρίσκονται σε ενεργεία. Για το κόστος τώρα της απασχόλησης ε, ε, όλων όσων είναι ανεργοί και δεν βρίσκονται σε ε, θέσεις εκπαίδευσης Υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες μελέτες από, τον, από, την, Διεθνή, από την Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, που λέει ότι ε, το κόστος αυτό είναι 44,8 ε, δις ευρώ. Αν τώρα δούμε τα συνολικά ποσά στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 86,4 δις ευρώ μεταξύ του 2014-2020. Άρα αυτά τα χρήματα δεν θα αρκέσουν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Ο στόχος της εγγύησης για, για την νεολαία είναι να αυξηθούν, να βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχολησιμότητας των νέων έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να παραμείνουν σε αυτήν. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου, θα πρέπει τα μέτρα αυτά ε, να ληφθούν εντός της ε, ε, εγγύησης των νέων. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφοράς των, και της ζήτησης των θέσεων εργασίας. Και βεβαίως θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι όσο περισσότερο απομακρυσμένοι, όσο πιο μακριά είναι από την αγορά εργασία τα άτομα, τόσο πιο πολύ κοστίζει να τους επανεντάξουμε σε αυτή. Μετά τους ε, ελέγχους του, δικαστικού, του συνεδρίου βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη που ήλεγξαν, οι παράμετροι δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη. Δηλαδή αυτή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των, της προσφοράς των δεξιοτήτων των υποψηφίων και της ζήτησης. Ε, βεβαίως ο πληθυσμός γυράσκει, αλλά πολλοί κόσμος ακόμη αναζητεί θέσεις εργασίας, οι νέοι κυρίως ε, προσπαθούν να μείνουν περισσότερο στην, στο πανεπιστήμιο, στην ε, ε, εκπαιδευτική ζωή και αναβάλουν το να μπουν στην αγορά εργασίας, ίσως όταν δουν ότι είναι καλύτερες οι συνθήκες στην αγορά εργασίας. Και πρέπει να πει κανεί ότι οι έλεγχοι του Ελεκτικού Συνεδρίου διαπιστώνουν ότι η προθεσμία αυτή των τεσσάρων μηνών στα ελεγχθέντα κράτη-μέλη δεν τηρήθηκε καν. Και επιπλέον έχουμε το ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την, ε, τον έλεγχο της κατάστασης των νέων εντός όλης αυτής της διαδικασίας. Τώρα, για, την, ε, για τον ορισμό. Βεβαίως ο ορισμός της ε, υψηλής, υψηλού επίπεδου εργασία παίζει σημαντικό ρόλο. Αν δούμε, ας πούμε, την Κροατία και τα δικά τους προγράμματα, λένε ότι η εγγύηση για τους νέους ε, βασίζεται σε, ή αφορά άτομα τα οποία γρήγορα μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα μέτρα. Και οι μακροχρόνια άνεργοι αργότερα θα μπορέσουν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Οπότε η... υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών που πρόσφατα έχασαν τη δουλειά τους και αυτών που είναι μακροχρόνια άνεργοι. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε υπόψη. Επίσης από τα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι τα άτομα που εποφελούνται από την εγγύηση των νέων είναι αυτά που έχουν τις καλύτερες δεξιότητες, την καλύτερη εκπαίδευση. Τα 7 κράτη που ελέγχθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο δείχνουν ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου σε ό,τι αφορά την εγγύηση των, για τους νέους, για την νεολαία. Παρόλα αυτά, οι συστάσεις του Συμβουλίου δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως και οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, κυρίως ό,τι αφορά αυτή την τετράμινη προθεσμία. Το 2014, 70% των θετικών των θετικών απαντήσεων καταγράφησαν. Το 2015 ο μέσος όρος βρισκόταν στο 59% δυστυχώς. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη-μέλη να, να εξεύρουν κάποιες στρατηγικές έτσι ώστε να μπορέσουν να καταγράψουν και να καταχωρήσουν τον πληθυσμό αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική με συγκεκριμένα μετρήσιμα στοιχεία, με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους ετησίως, με συγκεκριμένο τρόπο ε, συνέχισης των προγραμμάτων. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε την αγορά εργασίας και κυρίως αυτούς που βρίσκονται μακριά από αυτήν. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να έχουν και μια γενική εποπτεία του κόστους έτσι ώστε να μπορούν να, ε, να ε, καταγράψουν και το κόστος της ε, εγγύησης για, το, για την νεολαία και να καταρτήσουν τις προτεραιότητές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν κατά προτεραιότητα τα μέτρα αυτά που είναι τα πιο εύκολα, απο... που μπορούν να φέρουν τα πιο εύκολα αποτελέσματα. και για να συμπεριλάβουν τα άτομα που, μπορούν, ε, που το κόστος της συμπερίληψής τους είναι μικρότερο. Βεβαίως συμφωνούμε όλοι ότι η ε, μακροχρόνια άνεργοι βεβαίω χρειάζονται περισσότερη στήριξη, αλλά αυτή ίσω είναι μικρότερη ομάδα. Αν τώρα ε, πολλά, πολλοί πόροι πάνε σε μια μικρή ομάδα, ίσως ε, αυτό εμποδίσει κάποιους που έχουν καλύτερε ή περισσότερε δεξιότητε να βρουν μια θέση εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες προτάσεις για την προσφορά υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και για την αξιολόγηση αυτών. Τι σημαίνει δηλαδή υψηλής ποιότητας προσφορά? Μια προσφορά που θα αντικατοπτρίζει το προφίλ του υποψηφίου και θα καλύπτει και την ανάγκη της αγοράς. Μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας για την νεολαία ίσως είναι νωρίς να γίνει, αλλά κάποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Και βεβαίω η ε, απασχόληση των νέων είναι στον πυρήνα των αποφάσεων των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό σημείο. Και άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέους πόρους. Η ευελιξία δεν αρκεί. Όντως χρειαζόμαστε νέους πόρους. Ε, θα μπορούσε πολύ ώρα να μιλάω ακόμη, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα αυτό. Και ε, πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα όσα έγιναν το 2015. Το Κοινοβούλιο κατάφερε, όταν μιλούσαμε για τον προπολογισμό του για το 2016, μια περαιτέρω δέσμευση για την ε, ε, εγγύηση για την νεολαία. Τα κράτη-μέλη βεβαίω ήθελαν να αξιολογήσουν κατά την κατάσταση, δεν συμφωνούσαν απολύτω, η αξιολόγηση κράτησε ένα χρόνο και χάσαμε χρόνο τελικά. Γι' αυτό θέλω να πω ότι έχουμε τώρα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω ίσως για την χρήση στην εγγύηση για την νεολαία. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα στον κύριο Κόλμελ το λόγο, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, ευχαριστώ τον συνάδελφο Μάνκα για την διεξοδική του έκθεση. Αν δούμε τον τίτλο «Εγγύηση για την νεολαία», μιλούμε για καλή εκπαίδευση για τους νέους και καλές θέσει εργασία για τους νέους. Βεβαίω ε, θέλουμε να προχωρήσουμε ως προς αυτό. Παρόλα αυτά θα ήθελα να κάνω κάποια κριτική. Γιατί ήδη σήμερα βλέπουμε ότι ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Όσα ακούγονται ωραία δεν είναι πάντα ωραία. Έχουμε δει ότι για όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε προσωπικό, χρειαζόμαστε έλεγχο, εποπτεία, Αυτό τι είναι, γραφειοκρατία όμως. Και θέλω πάλι να θέσω ένα ερώτημα. Δεν θα ήταν σκόπιμο τέτοια μέτρα να τα ξανασκεφτούμε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει αρμοδιότητα για όλη την επικράτεια της Ένωσης. Κάνω τη διαφοροποίηση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες λόγω οικονομικής δυνατότητας και λόγω διοικητικής εμπειρίας δεν έχουν φτάσει, δεν έχουν προχωρήσει ε, τόσο πολύ όσο άλλες χώρες ίσως τις χώρες που είναι καινούριε, ας πούμε, θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε εμπειρία, ελάτε να σας βοηθήσουμε. Αλλά τώρα για την ε, Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, ε, όσο και να το σκεφτώ δεν μπορώ να φανταστώ πού ακριβώς υπάρχει η προστιθέμενη αξία για αυτές τις χώρες μέσω ενός μέτρου ευρωπαϊκού για την κατανομή πόρων. Ε, δεν χρειαζόμαστε τόσο περίπλοκες προσεγγίσεις. Δηλαδή δίνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας το δώσει πίσω. Είναι καλός λοιπόν ο τίτλος, αλλά πρέπει να σκεφτούμε αν όντως είναι σκόπιμα όλα αυτά. Και μια τελευταία φράση, Πρόεδρε, εδώ μιλούμε για τα συμπτώματα. Θα πρέπει να δούμε και την αιτία, την αιτία της υψηλής ανεργίας των νέων στην Ευρωζώνη. Το ευρώ είναι η αιτία. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Ça, c'est un diagnostic personnel. Πρόκειται για μια προσωπική διάγνωση αυτό που κάνατε κύριε Κόλμερ; Λοιπόν, τελειώσαμε με τους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα ομιλήσω την Πορτογαλική. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για την ε, παρουσίαση, τον κύριο Μάνκα. Όλοι θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα έχει αρμοδιότητα γιατί δεν μπορεί παρά να είναι ε, κοινός στόχος η μείωση της ανεργίας και η προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ιδιαίτερα στους νέους δυστυχώς η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή και είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράμματα. Το ίδιο κάνουν φυσικά και οι εθνικοί προϋπολογισμοί αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία θα έλεγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα. Ε, βλέπουμε στην παρούσα φάση να εμπλέκονται πάρα πολλοί νέοι ε, σε προγράμματα παρέμβασης στην Γεωργία, ένα παράδειγμα φέρνω την Γεωργία, για αρκετά χρόνια. Αυτά τα προγράμματα είναι πάντα προσωρινά και παραμένουν σε εκκρεμότητα οι σταδιοδρομίες τους και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να παρατείνεται χωρίς κανένα περιορισμό. Να δούμε λοιπόν, το ερώτημα είναι μέχρι σε ποια ηλικία μπορεί κανείς να διεκδικήσει, <clears throat> να είναι συγγνώμη, δικαιούχος κάποιων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την εγγύηση για τους νέους. Ε, Μέχρι τα 35, παραπάνω από τα 35, λιγότερο, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. είχαμε πει ότι εμείς θα πρέπει να πληκήσουμε τη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια με ένα δις 200 εκατομμύρια και θα πρέπει επίσης ε, να συνεισφέρουν και οι εθνικοί προϋπολογισμοί φυσικά. Εδώ το κοινωνικό ταμείο σαν παράδειγμα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο αλλά να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών προϋπολογισμών. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, λέει ο πρόεδρος έχουμε ένα πρόβλημα ανεργίας των νέων. Ε, είναι λίγες οι χώρες ε, οι οποίες δεν έχουν το πρόβλημα. Αυτό είναι οι χώρες που έχουν πολύ ισχυρά συστήματα μαθητείας. Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία αν ήταν μέλος. Γιατί να μην είμαστε λοιπόν σε θέματα μαθητείας και κατάρτισης πιο τολμηροί. Ε, δεν υπάρχει ένα καθεστώς μαθητείας εντωμεταξύ, κάθε χώρα έχει τα δικά της. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργήσει συνθήκες έτσι ώστε οι μαθητευόμενοι να μετακινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βλέπουν πώς δουλεύουν σε άλλες χώρες, εδώ το Εράσμος θα μπορούσε να τους καλύψει. Κύριε Μάνκα, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η συνταγή έτσι ώστε να καταστήσουμε τα κράτη-μέλη να ε, είναι πιο ικανά, εν πάση περιπτώσει, στο να προωθήσουν και την μαθητεία και την κατάρτιση για τους νέους και την κινητικότητα των μαθητευομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιο σχόλιο να κάνει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάνκα πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Φερνάντε. Το όριο ηλικία είναι διαφορετικό στα κράτη-μέλη. 25 χρόνια, 29 χρόνια, ανάλογα με το κράτος μέλος. Η ομάδα μου θα ζητήσει 30 χρόνια, εγώ στα 30 δηλαδή, να μπορούν να στηρίζονται οι νέοι και οι αναλύσεις επίσης ε, έχουν κάποιες αδυναμίες. Όταν σε ένα κράτος είναι το έτος ηλικίας 25 ε, και σε άλλα κράτη είναι 30, ε, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται κάποιο είδους ομοιογένεια. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Κάποιες χώρες έχουν λιγότερα προβλήματα με την ενεργεία των νέων ε, σε σχέση με άλλες. Η Δανία, ας πούμε, ε, κάνει training σε όλους τους ανέργους της, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα να βρουν μια νέα θέση εργασίας. Γι' αυτό η Δανία ανήκει στις ε, χώρες όπου και, και οι πολίτες ε, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και δεν αισθάνονται τόσο πολύ φόβο αν χάσουν τη δουλειά τους. Και αυτό έχει να κάνει με αυτή την προετοιμασία που τους γίνεται, με αυτό το training. Ελπίζω ότι όλες οι χώρες αργά ή γρήγορα θα μπορέσουν να βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται σίγουρα είναι μια ουσιαστική ανάλυση όλων των κρατών μελών. Ανάλυση της ανεργίας, έτσι ώστε να δούμε όλες τις ομάδες ανέργων και να δούμε πόσα χρήματα κοστίζει για να βοηθήσουμε όλες αυτές τις ομάδες ανέργων. Μια τέτοια ανάλυση λοιπόν είναι πραγματικά ε, επιγόντως απαραίτητη. Και τα χρήματα θα πρέπει βεβαίως να πάνε σε κάποιες ε, κατηγορίες. Ε, έχουμε λίγα χρήματα, άρα αυτά τα λίγα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουμε πολλά. Και ως προς αυτό χρειάζεται βιωσιμότητα και η βιωσιμότητα πάει χέρι-χέρι με την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη είναι το α και το ω δεν μπορούμε να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Το θέμα δεν είναι μόνο η αναργία ή η απασχόληση, το θέμα είναι πολιτικής φύσεως. Όταν κάποιος, ε, όταν ένας νέος είναι άνεργος, μπορούμε να τον χάσουμε και από πολιτική πλευρά. Μπορεί να παρατηθεί από τα πάντα και αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό υποστηρίζουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για να προχωρήσει το project αυτό. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε φρέσκα κονδύλια, νέα κονδύλια προς αυτό το πρόγραμμα. Να μην ανακυκλώνουμε μονίμως τα κονδύλια μας και να μην δίνουμε μόνο ad hoc λύσεις. Euh, Τώρα για το Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση έχουμε την περίπτωση της Φιλανδίας, ο κ. Σαβαρμά, Κοιτάξτε, είναι γνωστή η ιστορία, την έχετε ακούσει. Η Φιλανδία έχει καταθέσει για μια ακόμη φορά μια αίτηση για οικονομική συνεισφορά του συγκεκριμένου Ταμείου Προσαρμογής. 1247 απολύσεις της εταιρείας Microsoft Mobile και ε, συνεργαζομένων στην Φιλανδία. Συνολικό κόστος 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Το 60% θα καλύψει το Ταμείο Προσαρμογής, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια. Α, όπως είπα είναι παλιά και γνωστή ιστορία. Μειώνεται το κομμάτι της αγοράς της συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχουν ε, μειώσεις του της παρουσίας της επιχείρησης αυτής σε πολλές χώρες. Το 92,4% των δικαιούχων είναι από 25 μέχρι 34 ετών και έχουν υψηλό επίπεδο ειδίκευσης και μόρφωσης. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η επόμενη Πέμπτη, 13 Ιουλίου, 12η Μεσημβρινή. Και η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή μας στις 30 ή στις 31 Αυγούστου. Ευχαριστώ κύριο Σάβαρμα. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Ο κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για τον συνάδελφο Σέβαμα ένθρωμα για την έκθεσή του. Έχω πολλές αμφιβολίες για το σημείο αυτό. Το θέμα του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση νομίζω είναι ένα παράδειγμα αχρίαστων, αχρίαστης δαπάνης πόρων. Αν δούμε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλούμε συνέχεια για τη Microsoft, η οποία το 2016 είχε κέρδη 16 δις δολάρια. όπου έγιναν κάποιες συμφωνίες με την Φιλανδία, αγόρασε και μια εταιρεία, έφτιαξε τις θέσεις εργασίας, έκανε, πήρε πολλές επιδοτήσεις και αυτή η εταιρεία αποφασίζει να κλείσει την εταιρεία εκεί. Οπότε αυτό πραγματικά είναι ένας πολύ φτηνός τρόπος να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι πρέπει να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει μέτρα. Νομίζω ότι το πρώτο μέτρο θα ήταν η Φιλανδία με την Microsoft να καταλήξουν σε μια σκόπιμη διαδικασία, σε μια συμφωνία όπου θα συμμετέχει η Microsoft στην μετακπαίδευση αυτών των υπαλλήλων που θέλει να πωλήσει. Να τα μεταφέρουμε όλα στους ώμους της Ευρώπης νομίζω ότι είναι άσχημο και μάλιστα είναι λάθος με αυτό το ταμείο να, ε, και να ε, δημιουργούμε μέτρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ουσιαστικά για τα οποία δεν φταίει. Αυτά είναι λάθη των κρατών μελών και τα κρατημένη θα πρέπει να τα, να τα υπομισθούν. Αλλιώς δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε βεβαίω να επηρεάσουμε το πώ τα εθνικά κράτη θα κανονίζουν τα κέρδη του. Όμω, εάν ε, συμβαίνει αυτό να ζητούνται τέτοιες ε, ευκαιρίες από τα κράτη-μέλη, στήριξη από την Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει λόγω των tax ruling, των φορολογικών συμφωνιών. Είναι αρκετά ανόητα τα κράτη-μέλη ώστε να διαπράττουν ε, και να περνούν σε τέτοιες συμφωνίες. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της δημοσιονομικής συνοχής εδώ. Κύριε Σαβερμά, κοιτάξτε κύριε Κέλμελ, καταρχήν συμφωνούμε με τη βασική ιδέα που αναπτύξατε. Όμω στη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν μου αρέσει καθόλου που το λέω αυτό. Διότι το λέτε, θα πείτε επειδή είμαι Φινλανδός. Προσπαθώ να το προβάλλω. Αλλά ο λόγος που το λέω είναι επειδή προσωπικώς επισκέφτηκα τα εργοστάσια αυτά. Και είδα ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται τα ποσά. Πρέπει να πω ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα από τα, ένα από τους καλύτερους λόγους ε, και εκροής στα χρηματικά ποσά. Κατά τα άλλα, η Microsoft έχει αναλάβει όντως τις ευθύνες της. Εδώ, εντάξει, υπήρξε διαπραγμάτευση του κράτους με τη Microsoft, αλλά με λίγο χρήμα, 3,5 εκατομμύρια η πολιτική αξία θα είναι τεράστια, διότι το μήνυμα που στέλνουμε για το τι προσπαθούμε να κάνουμε και πόσο μας ενδιαφέρει το καλό των πολιτών μας θα είναι σημαντικό. Αξίζει τον κόπο, θεωρώ. Αξίζει να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαρβαμά, Κύριε Τάραν, θέλετε το λόγο σύντομα, γιατί έχουμε αργήσει. Ευχαριστώ, ναι, πολύ γρήγορα προς τον κύριο Κέλμελ να πω ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε εταιρείε όπως η Microsoft έχουμε πολύ καλούς ε, συνεργάτες όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πληρώνουν τεράστιες ε, άδειες ε, τέλη αδειών για το λογισμικό στη Microsoft. χωρίς καμία συμφωνία για δωρεάν λογισμικό από άλλες εταιρείες. Έγινε μια δεκαετή συμφωνία και δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη που θα έπρεπε να δακτυλοδείχνουμε εδώ. Μην τους ε, θεωρούμε μόνο εκείνους πολύ υποχωρητικούς απέναντι των πολυεθνικών. απέναντι στις πολυεθνικές. Ευχαριστώ. Ας ε, το αφήσουμε εδώ το θέμα και να περάσουμε τώρα σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμήνης. Το ιστορικό για το πώς θα προχωρήσουμε στην εξέταση του θέματος. Μία ώρα πρέπει να αφιερώσουμε αυτό που θα μας φτάσει περίπου στις 12.40. Θα ζητήσω από όλους να μας συγχωρήσουν καθότι καθιστορήσαμε και θα ζητήσω συγγνώμη και από τους μεταφραστές. Από την Επιτροπή ο υπεύθυνο θα μας κάνει μια παρουσίαση δεκάλεπτη ε, επικεντρωνόμενος στις βασικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμήνης. Την παρουσίαση αυτή θα ακολουθήσει μια σειρά από ερωταπαντήσεις. Ο κύριος Αλέξη, ο υπεύθυνο των θέματων αμήνης στη DigiGrow, που η DG Grow να υπεύθυνη στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα δώσει ενδεχομένω απάντηση. Επίσης έχουν προσκληθεί τα μέλη των Επιτροπών Ήτρε, ΣΕΝΤΕ και ΑΦΕΤ και ευχαριστώ όσου ήρθαν εδώ και τους εύχομαι ε, το καλώ όρισε. Οι συντονιστέ τη 29 Ιουνίου ε, παρακολούθησαν το θέμα τη επιμηχανική ανάπτυξη για την άμυνα και ο εισηγητή του, του ΕΛΚ ε, θα πρέπει να τοποθετηθεί. Με εισηγητή μάλλον του ΕΛΚ θα πρέπει να τοποθετηθεί, δεν τον ξέρουμε ακόμα, θα μα πει ο κύριο Φερνάντε να το ξέρει. Δίνω το λόγο στον υπεύθυνο τη Επιτροπή για μια δεκάλεπτη παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να παραμείνω εντό των ορίων. Θα ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμήνη συνολικά και μετά πολύ γρήγορα θα έρθω στην ε, πρόταση επιτάπητος που είναι το βασικό σημείο που μας ενδιαφέρει σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας αποτελείται από δύο διαφορετικά παράθυρα θηρίδες. Πρώτα απ' όλα τη θηρίδα της έρευνας, η οποία χρηματοδοτεί συνεργατικά προγράμματα έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το δεύτερο είναι το παράθυρο δυνατότητας, θηρίδα δυνατότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού για να αυξηθεί το σύνολο των ε, επενδύσεων στα αμυντικά προγράμματα και για να μειωθεί ο κατακαιρματισμός του κλάδου που αυτή τη στιγμή είναι οργανωμένος εντελώς σε εθνική βάση. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο θηρίδες, αυτά τα δύο παράθυρα και έχουμε και χρονικές θηρίδες. Έχουμε δηλαδή το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από τη μια και το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την άλλη. Τέσσερα διαφορετικά ε, μπλοκ σύνολα δαπανών που μας ενδιαφέρουν εδώ. Στο παράθυρο της έρευνας έχουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έρευνα για την άμυνα, όπου προβλέπαμε 90 εκατομμύρια σε μια τριετία, 2017, 2018, 2019. Δεν θα τα αναπτύξω αυτά με λεπτομέρειες σήμερα. Στο παράθυρο της επένδυσης για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να προδικάσουμε βεβαίω τι αποφάσει που θα ληφθούν για το ερχόμενο που Όμω, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προτείνει ένα πρόγραμμα έρευνα για την άμυνα που να αξίζει συνολικά 500 εκατομμύρια ετησίως. Ξεχωριστά και επιπλέον από το νορίζοντα 2020. Αυτά ως προς την έρευνα και τη θηρίδα της. Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και το σχετικό παράθυρο θηρίδα. Εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συνδυάσουμε εθνικές συνεισφορές που θα συγκεντρωθούν και αυτά να συμπληρωθούν από στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να έχουμε 80% της συγκέντρωσης των εθνικών συνεισφορών και 20% στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Προτείνουμε ο λόγος αυτός να ισχύει και για το τωρινό πουδουπού και για το μελλοντικό. Για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό μετά το 2020, η ιδέα είναι να κινητοποιήσουμε συνολικά 5 δις ετησίως με τον λόγο 20 προς 80, δηλαδή 4 δις από τις εθνικές συνεισφορές, τα οποία να είναι συγκεντρωμένα, και 1 δις από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ετησίως. Τώρα, να έρθω στην πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Το, τη θηρίδα δυνατοτήτων για το τωρινόπουδο που το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες εβδομάδες έκανε μια πρόταση να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή κό πρόγραμμα ε, βιομηχανικής ανάπτυξης της άμυνας. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 500 εκατομμύρια ευρώ χαρτοφυλάκια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για το 2019-2020. 500 εκατομμύρια δηλαδή για το τωρινό που και αυτό συντεριάζει με τη συνολική μας προσέγγιση το λόγο του 80 προ 20%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή προτείνει 2 δις να είναι οι συνεισφορές των ε, κρατών μελών και συνολικά θα έχουμε 2,5 δις από το τωρινό ποδοπό για την Ευρωπαϊκή Συνεισφορά. Ως προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση αυτών των 500 εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μείγμα χρηματοδότησης, 75% για την ε, επαναδίπλωση και 25% φρέσκο χρήμα. Τα ε, ποσοστά αυτά θα είναι οικία τα μέλη της Επιτροπής σας, διότι συνάδουν με άλλες προτάσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια για την ε, χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων στον ε, τίτλο 1α. Ε, τον ίδιο λόγο είχαμε προτείνει για το S1, για το SI2 και πιο πρόσφατα προτείναμε τον ίδιο λόγο 75 προς 25 για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού ε, Σώματος Αλληλεγγύης. Άρα, η πρόταση εδώ για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Άμυνας και ε, Βιομηχανικής Ανάπτυξης ακολουθεί το λόγο 75 προς 25%. Εάν συνολικά έχουμε τα 500 εκατομμύρια όπως προτείναμε, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 25% φρέσκο χρήμα, δηλαδή 125 εκατομμύρια από το περιθώριο που δεν έχει αποδοθεί στο 1α 2019 και 2020 και 375 εκατομμύρια ε, 75%. Redeployment. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 375, 375 εκατομμύρια προτείνει το εξή. Το πρώτο που θέλαμε να κάνουμε προφανώς, είναι να σεβαστούμε την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πουδουπού. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου προτείνει top-up για προγράμματα όπως το Ορίζοντας 2020, το ΣΕΦ των μεταφορών, το Erasmus ΣΥΝ και το κόσμο. Δηλαδή, για μας όλα αυτά ήταν τα επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο αυτής της πρότασης, διότι δεν θα ήταν λογικό να τα αγγίξουμε αυτά και να πάρουμε μη χρησιμοποιημένα ποσά από εκεί, αφού το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ήθελαν να τονώσουν τα προγράμματα αυτά στο τωρινό ποδοπού. Αυτά τα σημαντικά λοιπόν προγράμματα του τίτλου 1α δεν έπρεπε να τα αγγίξουμε. Αυτό βεβαίω περιόρισε το περιθώριο ε, λιγμού για να βρούμε εμεί ποσά μη χρησιμοποιημένα να τα αξιοποιήσουμε και κάνουμε την εξή πρόταση προ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα προτείνουμε επαναχρησιμοποίηση 120 εκατομμυρίων από τις δωρεές του ΣΕΦ για την ενέργεια. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, ακαθόδε ζήτημα για την Επιτροπή σας. Επίσης υπό το φως των διαπραγματεύσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη για το FSI 2 εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει επαναχρησιμοποίηση μεταξύ άλλων από το ΣΕΦ ενέργειας έτσι κι αλλιώ, αλλά θέλω να καταστήσω σαφές ότι κατά την άποψη της Επιτροπής υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του σημείου υλοποίηση και εφαρμογή εκτέλεση μάλλον του ΣΕΦ για την ενέργεια και του ΣΕΦ για τι μεταφορέ. Και αυτό όχι μόνο για λόγου ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά και για λόγους ε, συμφυής με το ε, στάδιο υλοποίηση των προγραμμάτων. Να μην αγγίξουμε το ΣΕΦ μεταφορών προτείνουμε, αλλά για το ΣΕΦ της ενέργειας, κατά πρώτον, στο ΣΕΦ της ενέργειας, τα χαρτοφυλάκια θα ευξηθούν ούτως ή άλλως σημαντικώς, όπως έγινε τα τελευταία χρόνια του Πουδουπού, και αφού ληφθεί υπόψη η επαναχρησιμοποίηση που προτείνεται για το σαι και αφού ληφθεί υπόψη και επαναχρησιμοποίηση που ε, προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άμυνας και πάλι θα υπάρξει αύξηση 36% στο ΣΕΦ στο χαρτοφυλάκιό του μεταξύ του 2018 και του 2019 και μετά κι άλλη αύξηση 21% μεταξύ 2019 και 2020. Οπότε, προφανώς, κατά τη δική μας την κρίση, υπάρχει περιθώριο να ε, υποβάλουμε προτάσεις για να πάρουμε ποσά, σημαντικά ποσά στο μέλλον από το ΣΕΦ ενέργειας. Είναι γεγονός, Δυστυχώ ίσως, ότι σε αυτή τη φάση το πώς προχωρούν τα προγράμματα και οι δωρεές τους για το ΣΕΦ της ενέργειας δεν έχει δείξει με όριμο τρόπο ότι προχωρά σωστά. Πάνω από το ίμιση των προτάσεων ε, για, στα πλαίσια του πουδου που προ στιγμή δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Ε, υπάρχει ελλειπή υποβολή έργων ε, σε σχέση με το σεφ τη μεταφοράς και αν δούμε τα χαρτοφυλάκια του 2019 μέσω των πολυετών ε, προμηθειών μόνο 25% των χαρτοφυλακίων αυτών των ετών έχουν αναλυφθεί και έχουν καλυφθεί. Αυτό επηρεάζει το ΣΕΦ ενέργειας, ενώ στο ΣΕΦ μεταφορών μόνο 19% έχουμε ήδη κρατήσεις, για να το πω έτσι, για τα χαρτοφυλάκια το 2019-2020. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το ΣΕΦ ενέργειας υπάρχει περιθώριο για την επαναχρησιμοποίηση και δεν θα προκαλέσει ολιγορίες, καθυστερήσεις ή αναβολές των έργων της ενέργειας που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται. Το δεύτερο στοιχείο της χρηματοδότησης, τα 25 εκατομμύρια, θα είναι από το ΣΕΦ του ICP. Ε, εδώ υπάρχει συνέργεια πολιτική, διότι ήδη χρηματοδοτούνται έργα στα, στο χώρο της κυβερνοασφάλειας λόγου χάρη. Υπάρχουν και διαδικασίε για την υποβολή ενδιαφέροντο ε, για ποσό 21 εκατομμυρίου από το 2014 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτάζει να δημιουργηθούν σχέσει συνεργασία μεταξύ τη κυβερνοασφάλεια και ε, τη άμυνα γενικότερα. Υπάρχει λοιπόν πολιτική ε, λογική στο να πάρουμε αυτά τα 25, αυτά τα 25 εκατομμύρια ως επαναχρησιμοποίηση από εκεί. Τώρα, κατά τα άλλα, για το ποσοστό αυτό θα έχουμε χρηματοδότηση από τα έργα μεγάλη κλίμακας Γαλιλαίο, Κοπέρνικους και Ίτερ για ένα συνολικό ποσό 230 εκατομμυρίων και για τα τρία μαζί. Κατά πρώτον από το Γαλιλαίο προτείνουμε να χρησιμοποιήσει 135 εκατομμύρια. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εφικτό, διότι τον Γαλιλαίο έχει σημαντικά ποσά εσόδων ε, προ ειδικό σκοπό, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη για... με πολύ καλό τρόπο, αλλά υπάρχει και ένα περιθώριο ελιγμού εδώ. Τα ειδικά αυτά έσοδα για ε, ειδικό σκοπό προέρχονται από την Νορβηγία και την Ελβετία, που συμβάλλουν σημαντικά στον Καλιλαίο κάθε χρόνο. Επιπλέον από τα ποσά που έχουν προγραμματιστεί στο Πουδουπού. Δεδομένων λοιπόν αυτών των ποσών, των assigned revenues, των εσόδων για ειδικό σκοπό, πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με την επαναχρησιμοποίηση των 135 εκατομμυρίων, τα οποία εκπροσωπούν 9,9% περίπου νομίζω από το συνολικό χαρτοφυλάκιο του Γαλιλαίου. Το ίδιο και για το Κοπέρνικους, 15 εκατομμύρια. Νομίζω μπορούμε να τα πάρουμε από τα ειδικά έσοδα, τα έσοδα για ειδικό σκοπό και τα υπόλοιπα προτείνουμε να έρχονται από το ΙΤΕΡ, προτείνουμε ένα ποσό 80 εκατομμυρίων. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν ήταν εύκολο να τα βρούμε. είμαστε οριακά στην επαναχρησιμοποίηση εδώ για το πρόγραμμα αυτό στο τωρινό, στο τρέχον από το που, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας νέας πρότασης που έγινε από τη διεθνή οργάνωση του ΙΤΕΡ για την περίοδο προγραμματισμού 2017-2020 και ελπίζουμε ότι το χρηματικό αυτό ποσό μπορούμε να το πάρουμε για την άμενα χωρίς να εκθέσουμε τις υποχρεώσεις της Ένωσης ενώπιον της Διεθνούς Οργάνωσης για το ΙΤΕΡ. Θα σταματήσω εδώ για να μείνω εντό των χρονικών πλαισίων και μαζί με τον συνάδελφο από την DG Grow είμαστε έτοιμοι για να απαντήσουμε στι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Φερνάντες. Το θέμα είναι τι περιθώρια έχουμε στη συγκεκριμένη στιγμή. Το δεύτερο ερώτημα είναι πότε επιτέλους τα όργανα θα σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει το λεγόμενο «Pacta sunt servanda». Εγώ υπενθυμίζω ότι έχουμε πάρει αρκετά χρήματα από άλλα μέσα, όπως επίσης και από το Horizon 2020, μεγάλα ποσοστά, για να χρηματοδοτήσουμε το Στρατηγικό Ταμείο 1. Τώρα η πρόταση της Επιτροπής και το Συμβούλιο είναι επίσης να πάρουν ξανά χρήματα και για το ε, FC2, το Στρατηγικό Ταμείο Υπαριθμών 2 και τώρα πάλι και για την άμυνα. Εντάξει, είναι νέα προτεραιότητα, αλλά ποια είναι η λογική. Είναι σαφές ότι οι νέες προτεραιότητες θα πρέπει να τύχουν δημοσιονομικής κάλυψης μέσω μιας συγκεκριμένης πίστοσης. Συνεπώς απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω, γιατί δεν το κατάλαβα πολύ καλά, αν τα 147 εκατομμύρια είναι, από πού ακριβώς προέρχονται. Ε, ε, προέρχονται από επιδοτήσεις, από επιχορηγήσεις ή προέρχονται από άλλου είδους χρηματοδοτικά μέσα. Ελπίζω η απάντηση η οποία θα μου δοθεί να μας διευκρινίζει το περιθώριο το οποίο έχουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα εξηγηθεί και γιατί προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από το περιθώριο αυτό μόνο το ποσό των 120 εκατομμυρίων. Στην ουσία αυτό το οποίο επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να πολλαπλασιαστεί ο προϋπολογισμός ένα δις επιπλέον από τη μία λένε στη Γαλλία, το παίρνεις όμως από τη μία τσέπη και το βάζεις στην άλλη και στην ουσία ναι μεν πολλαπλασιάζεις τους αριθμούς, στο τέλος όμως οι αριθμοί παραμένουν οι ίδιοι. Στην ουσία το μόνο το οποίο κάνουμε συνάδελφοι είναι να περικόπτουμε τα ισχύοντα προγράμματα, τα οποία είναι σημαντικά προγράμματα και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πρέπει λοιπόν, εφόσον θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις προτεραιότητές μας τις νέες, να κάνουμε μία επιπλέον προσπάθεια. Θα πρέπει ε, να είμαστε βέβαιοι το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι συνεισφορές οι εθνικές. Με ποιο τρόπο θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τύχει σωστής απάντηση. Η κυρία Γουαρδιαζάμπαλ, ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος Νομίζω ότι θα συμφωνήσω άλλωστε σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία είπε ο Χουάν Μανουέλ Φερνάντες. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε πει χίλιες φορές μέχρι τώρα ότι για νέες πολιτικές χρειάζονται νέες πιστώσεις, νέες χρηματοδοτήσεις. Τι νόημα έχει εμείς να καθορίζουμε προτεραιότητες, να φτιάχνουμε προγράμματα και τις προτεραιότητες αυτές να μην μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε και να εξαφανίζονται. Με εκπλήσει λοιπόν, δηλαδή τώρα δεν με εκπλήσει και πολύ εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην λέμε τα ίδια. Εμείς έχουμε θέσει κάποιες προτεραιότητες, δυστυχώς δεν ε, καλύπτονται στον προϋπολογισμό ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια μικρή εσωτερική κουζίνα για να καλύψει αλλά μόνο περιφερειακά ε, τους δικούς μας στόχους και τις δικές μας προτεραιότητες και μόνο στόχος ουσιαστικός είναι η κάλυψη των αναγκών του στρατηγικού ταμείου. Τι νόημα έχουν και οι τριμερείς διάλογοι, δεν έχει νόημα να φέρνουμε από την ενέργεια, να δίνουμε αλλού, να προσπαθούμε να κινηθούμε με τις προκαθορισμένες επιδοτήσεις, τα ειδικά έσοδα έτσι δεν υπάρχει λύση. Καλά τα είπατε, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Τα ουσιώδη νομίζω υπόθηκαν. Και επειδή πρέπει να εξοικονομήσουμε για χρόνο, δεν θέλω το λόγο. Ευχαριστούμε, κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν είμαι εγώ για την ομάδα μου αλλά θα συμπαραταχθώ με τον κύριο Φερνάντε τι ίδιε ερωτήσει έχω και εγώ. Ευχαριστούμε κύριο Στάραντ. Αγαστή ε, συνεργασία. Θα σα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Φερνάντε. Monsieur Finch qui remplace Monsieur Arnott. Thank you, Mr. Chairman. Ε, στη θέση του κυρίου κύριο Φίντ. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω για τα 5 δι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Βασίζεται στην εικασία ότι θα έχετε ακόμα τι συνεισφορέ του Ηνωμένου Βασιλείου στην ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ε, αν όχι, με τα προγράμματα που θα περικοπούν, τι θα γίνει. Τα υπόλοιπα κάτι μέλη θα βάλουν περισσότερο χρήμα Merci. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε αφήνοντα τους συντονιστέ ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσει και μια ερώτηση. Πρώτη παρατήρηση. Είμαστε βέβαιοι για το τι θα κάνουμε με το ΣΕΦ, διότι οι συζητήσεις ε, κάνουμε εδώ και χρόνια. Και λέγαμε αν είναι απαραίτητο ή όχι το πρόγραμμα αυτό. Τώρα του πειράζουμε το αποθεματικό, όπως είπε και ο Ζωζέ. Θα προκύψει θέμα εδώ. Διότι αν κόβουμε και κόβουμε, αρχίζει πάλι να τίθεται το ερώτημα αν χρειάζεται ή όχι αυτό το πρόγραμμα. Εκτό και αν πολιτική μα. Δεύτερη παρατήρηση. Να υπογραμμίσω απλώ ότι έχουμε top-up στην ενδιάμεση αναθεώρηση και υπάρχει και υποσημείωση τη θέση του Κοινοβουλίου εδώ, ότι αυτό δεν μειώνει την ε, εποπτεία του Κοινοβουλίου για τον ετήσιο προπολογισμό, είναι ένα τμήμα στο οποίο θέση μπορεί να πάρει και το Κοινοβούλιο για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ανοίγει συζήτηση και δεν είναι θέμα απλώ δημοσιονομικό. Είναι κάτι που προτινόταν και είχαμε πει εντάξει, αλλά θα το δούμε και στην ετήσια διαδικασία του προπολογισμού. Το αληθινό ερώτημα είναι το ερώτημα του μελλοντικού ποδοπού. Εάν σήμερα αποφασίσουμε ότι αυτές είναι οι προτεραιότητες, τι συνέπειες θα έχει αυτό για το μέλλον. φρέσκο χρήμα που θα βρεθεί από τον προπολογισμό. Προφανώ δεν θα βρεθεί, διότι αν ανοίξουμε τώρα το θέμα τη μεθοδολογία, ουσιαστικά καθορίζουμε και το μέλλον. Είναι κάτι το προσωρινό δηλαδή αυτό, είναι μια μόνιμη λύση. Η πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κάνει την άμυνα προτεραιότητα και για το μέλλον καταλαβαίνω ότι είναι ένα δι ετησίω από το 2021. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Αν επιτρέπουμε να πηγαίνουν τα χρήματα από εδώ και από εκεί, ε, δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε παρόμοια καλή ε, εμπειρία στη Γερμανία. Γιατί βάζουμε στη χρήματα σε μια ανατομία που δεν έχουμε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Στην άμυνα δεν έχουμε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Θέλουμε να προχωρήσουμε με τα σημαντικά θέματα βεβαίως, αλλά αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι αυτά τα νέα θέματα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις υπάρχουσες προτεραιότητες. Νομίζω ότι κάνουμε τεράστιο λάθος αν μπούμε σε αυτή την ατραπό. Και νομίζω ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Αν θέλουμε νέε προτεραιότητε, νέα καθήκοντα, για τα οποία δεν έχουμε καν ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, εκεί θα πρέπει να υπάρχει νέο χρήμα στο Ταμείο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιο μεγάλο λάθο, να βάλουμε νέε προτεραιότητε, τι οποίε θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε με υπάρχοντα κονδύλια, ενώ δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαγιέρ. Δεν ξέρω και από πού να αρχίσω. Ε, γιατί εκπλήσωμαι, θυμώνω ταυτόχρονα. Θυμώνω καταρχάς για το ότι αυτή η Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια Μιλάει για την ενίσχυση των κονδυλίων για κάποιους τομείς. Εμείς από το, από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν πάντα λαμβάνουμε απάντηση γιατί δεν είναι όλα αυτά χρηματοδοτήσιμα. Τώρα, το θέμα της ασφάλειας και της ε, άμυνας έχει πάρει μεγαλύτερη συζήτηση στην, στο Συμβούλιο και άρα υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου το Συμβούλιο είναι σε θέση να συμφωνήσει. Η πραγματικότητα πραγματικά είναι ελλειπής και αυτό με οργίζει. Γιατί αυτή η ιεραρχία στόχων, πραγμάτων που είναι για κάποιον σημαντικά και που μπορεί να κάνει τα πάντα και άλλων πραγμάτων που δεν είναι τόσο σημαντικά και που πάντα καταραίουν, ε, είναι συγκλονιστικό να συμβαίνει και εμένα με οργίζει. Οπότε, συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφο Γκρέσλε. Πριν ξεκινήσουμε να ρίχνουμε λεφτά από εδώ και από εκεί, Α συζητήσουμε για κάτι άλλο. Α συζητήσουμε για τι προτεραιότητε που έχει το Κοινοβούλιο και για, την για τι οποίε υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν και λεφτά. Α δούμε το θέμα τη συναπόφαση. Τέσσερα δι θα έρθουν, λέει, από τα κράτη-μέλη, από αυτή τη θηρίδα δυνατοτήτων. Ε, Προβλέπετε ότι αυτός εδώ ο οίκος σε αυτή την λαθασμένη χρηματοδότηση από, με τα 4, κράτη, δις από τα κράτη-μέλη και 1 δις από το δικό μας τον Κορβανά θα μπορέσει να επηρεάσει κάπως τα πράγματα. Θα μπορέσουμε δηλαδή εμείς να έχουμε κάποιο λόγο. Αν δεν το αποφασίσουμε αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητήσουμε ούτε για ένα απλό επιπλέον. Γιατί ένα δις το οποίο δεν ξέρουμε αν θα έρθει από τα κράτη-μέλη στα επόμενη ενδιάμεσο πολιετές πλαίσιο, θα πούνε, ναι, τα κράτη-μέλη, ναι, αλλά η, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εδώ πέρα ε, αρμοδιότητα, δεν μπορεί να παρέμβει και θα καταρρεύσουν πάλι τα πάντα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα και γιατί, για τούτη την Επιτροπή νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικά. Πριν να έχουμε και για τη διαδικασία αλλά και για την ουσία πληροφορίες, αν εγώ δεν διαβάσω τίποτα σχετικά, δεν έχω καμία διάθεση να κάτσω να συζητήσω για το ποια είναι τα κονδύλια που θα πάνε σε ποιο πρόγραμμα και πώς θα γίνουν όλα αυτά. Και επειδή ακριβώς έχουμε προτεραιότητες για τις οποίες πάντα λαμβάνονται αποφάσεις, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ψηλά στις δικές μου προτεραιότητες αυτά τα 500 εκατομμύρια και τα 375 και τα 125 να τα ξανασυζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει η Κομισιόν. Thank you very much for giving me the word. My name is Anna. Ε, προέρχομαι από την Επιτροπή ΑΦΕΤ και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο μόλις τώρα είπε ο Γκάγερ. Έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με μία νέα αρμοδιότητα. Το πλαίσιο το δημοσιονομικό το οποίο έχει διαμορφωθεί ε, επηρεάζει φυσικά και τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα είναι ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει σαν παράδειγμα με το καθεστώς ε, απαγόρευσης εξαγωγών σε ορισμένα είδη τέτοιες στρατιωτικά ειδητής χρήσεως και δεν ξέρω αν θα παραμείνει η ονομασία ευρωπαϊκής εξαγωγικής πολιτικής. Ξέρω ότι και ξέρετε κι εσείς ότι τα περισσότερα όπλα ελεύθερα εξάγονται, απαγορεύεται ε, υποτίθεται η εξαγωγή ε, άλλων μέσων, ε, βασανιστήριων κτλ. Το θέμα είναι λοιπόν να προσπαθήσουμε να μην χάσουμε τον έλεγχο της υπόθεσης και κυρίως σε ό,τι μας αφορά να μην χάσουμε τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Ο κύριος Σάρμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία σαφέστερη διάκριση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Πρώτο, αν έχουμε να κάνουμε με φρέσκο χρήμα και αν ναι, ποιος το δίνει αυτό το φρέσκο χρήμα. Και το δεύτερο πράγμα είναι το γιατί θα πρέπει να το έχουμε αυτό. Υπάρχουν ε, κάποιες, ε, κάποιοι δισταγμοί, κάποιοι έχουν φύγει ήδη που είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, αλλά ακούγονται φωνές και αρκετά επιθετικές σε σχέση με τις προτάσεις αυτές όπως του κ. Γκάια. Προφανώς και θα πρέπει να είναι φρέσκο το χρήμα, επιπλέον χρήμα, γιατί θα ωφεληθούν τα ίδια τα κράτη-μέλη, τα οποία χάνουν τεράστια ποσά στον τομέα των δαπανών των αμυντικών. Τα ποσά αυτά τα χάνουν διότι ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη-μέλη είναι αναποτελεσματικός. Αν δείτε τα ποσά τα οποία δαπανώνται στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένε Πολιτείες, κατανοείτε ότι είναι ε, ε, φρικτό αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη. Δεν είμαστε ηγέτες βιομηχανική δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας, δεν παράγουμε τα επιθυμητά όπλα. Πραγματικά ο λόγος ανάμεσα στα, στην αποτελεσματικότητα τη δική μας και των Αμερικανών είναι ένα προς πέντε. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε σωστά τα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρουμε ότι για το πολιετές δημοσιονομικό μετά το 20, δύο είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν. Το ένα είναι το μεταναστευτικό και το άλλο είναι τα θέματα της ασφάλειας. Ας δούμε λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τις δυνατότητές μας και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και φυσικά τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς γιατί άμεσα οι εθνικοί προϋπολογισμοί, δηλαδή οι ίδιες οι χώρες είναι αυτές που θα ωφεληθούν. Και υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα το οποίο υπερκαλύπτει τα υπόλοιπα. Αν θέλετε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας μετά το 2020. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολιτικά μια βασική προτεραιότητα. Οπότε γιατί να μην προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή όντας περισσότερο αποτελεσματική. δεν είναι κάτι το οποίο σαφώς ανήκει στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κοινέ προσπάθειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν καλύτερη χρήση των διαθεσίμων πόρων και κυρίως συνδυασμένη χρήση των διαθεσίμων πόρων. Ε, λοιπόν δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Είναι σαφές ότι οι προτάσεις αυτές συνιστούν μια ουσιαστική καινοτομία η Ευρώπη της άμυνας. Αλλά μιας και είναι τόσο σημαντική η πρωτοβουλία αυτή, δεν θα πρέπει η Επιτροπή να είναι λίγο πιο πραγματιστική και να ζητήσει να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερα τις μελλοντικές εξελίξεις ε, στον τομέα της ε, άμυνας δεν μπορούμε να έχουμε 17 τύπους ε, τεθωρακισμένων πρώτης γραμμής. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα αναχαιτιστικά αεροσκάφη που υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση ιστορικής αναποτελεσματικότητας. Αν θέλουμε η Ευρώπη να καταστεί μια πραγματική διεθνής ε, δύναμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό. Ξέρω ότι η μέθοδος που ακολουθείτε τελευταία είναι το να βάζει κανείς το πόδι στην πόρτα για να μην κλείζει και να ελπίζει ότι από εκεί και πέρα θα ανοίξει η πόρτα διάπλατα. Δεν είναι έτσι το θέμα όμως. Νομίζω ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να παρουσιάσει το τι είναι καλό για αυτήν. Δυσκολεύεται να βοηθήσει την κοινή της γνώμη να την στηρίξει. Έχουμε λοιπόν δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ιουρελ για τον προϋπολογισμό και τον κύριο Αλεξή για την Γενική Διεύθυνση Γκρό. Ο κύριος Ιουρελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για αυτό που θεωρώ ότι εκφράζει γενική στήριξη για την άμυνα αυτή καθεαυτή. Ωστόσο, ταυτόχρονα ε, σημειώνω και τις πολλές επικρίσεις για το χρηματοδοτικό μείγμα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί του οποίου φυσικά πρέπει να τοποθετηθούμε και σημειώνουμε τις απόψεις θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ειδικότερε ερωτήσεις κυρίως του κυρίου Φερνάντες. Πρώτη ερώτηση ήταν πόσο περιθώριο έχουμε ακόμη υπό το 1α σε αυτή τη φάση. Στο στην περίοδο προγραμματισμού μαζί με το σχέδιο προπολογισμού 2018, τα μη αποδιδούμενα περιθώρια για το 2019 και 2020 συνδυασμένα δίνουν 660 εκατομμύρια ευρώ. Εάν αφαιρέσουμε τα 125 εκατομμύρια που περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση της άμυνας και επίσης διαφυλάξουμε ένα ελάχιστο περιθώριο για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις του Ευρωκοινοβουλίου και αναφερέσουμε και άλλα 100 ή 50 εκατομμύρια ετησίως που είναι το ελάχιστο όριο, τότε τα 660 εκατομμύρια θα φτάσουν τα 435. 171 ε, το 2019 και 264 το 2020. Η επόμενη ερώτηση του κ. Φερνάντε είναι εφόσον υπάρχουν αυτά τα περιθώρια, γιατί δεν τα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νομίζω η απάντησή μου θα είναι και αναμενόμενη είναι θέμα κατά την άποψή μας σύνεσης. Σε αυτή τη φάση είμαστε ακριβώς στο σημείο καμπή στη μέση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε 3,5 έτη πίσω μας και 3,5 έτη μπροστά μας. Ήδη έχουμε δει μεγάλο αριθμό νέων εξελίξεων στο 1α, όπου προτάσεις με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, υπευλήθησαν. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές εξελίξεις τα επόμενα 3,5 χρόνια, οπότε κατά την άποψή μας Αναγνωρίζουμε μεν ότι κάποιο ποσό φρέσκου χρήματος χρειάζεται, γι' αυτό και προτείναμε τα 125 εκατομμύρια, όμως ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, 3,5 χρόνια πριν το τέλος του Πουδουπού, συνετό θα ήτο να διατηρήσουμε τα 435 εκατομμύρια ε, ανέπαθα για τις ενδεχόμενες μελλοντικές εξελίξεις. Ναι, αν μου επιτρέπετε όμως, ο κύριος Φερνάντες έχει μια σύντομη υπερώτηση. Ναι, για αυτό το σημείο. Γιατί μιλάτε για τον τίτλο 1α και το περιθώριο εκεί. Έχουμε ένα συνολικό περιθώριο και το ερώτημά μου δεν είναι μόνον πόσο έχουμε στο 1α περιθώριο, αλλά από όλα τα κεφάλαια και τίτλους τι περιθώριο έχουμε. Για το 1B παραδείγματος χάρη, για το 1β. Μα ακριβώς για τον ΠΗ δεν έχουμε περιθώριο. Τα περιθώρια στους υπόλοιπους τίτλους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 1α. Αυτό που υπάρχει, εν, ίσως αυτό εννοεί ο κύριος Φερνάντες, είναι το γενικό περιθώριο πιστώσεων, τα ειδικά εργαλεία. Ναι, αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η επιπλέον δυνατότητα. Ήδη χρησιμοποιήσαμε το γενικό περιθώριο της πιστώσης με τρόπο πολύ σημαντικό για την ε, χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Δεν προτείναμε να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί και αυτή η πρόταση. Πάλι το ίδιο. Για λόγους σύνεσης. Σύνεσης. Όμως είναι σαφές ότι η δυνατότητα υπάρχει. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Πόσο είναι το περιθώριο αυτή τη στιγμή από το γενικό περιθώριο που λέτε. Πόσο είναι. Πρέπει να απαντήσω γραπτός. Δεν έχω τον αριθμό εδώ. Θέλω να μου το πείτε. Θέλω να μου το πείτε γιατί η ένδειξή μου είναι ότι είναι πάνω από 2,6 δις ευρώ. Και είμαι βέβαιος ότι δεν τα χρησιμοποιήσατε τα 2,6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του Πουδοπού Θα το κοιτάξω, να το επιβεβαιώσω και θα το επαληθεύσω γραπτός. Θα το κάνω αμέσως, αμέσως σήμερα κιόλας. Όμως, να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση, το γενικό περιθώριο των πιστώσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τα κεφάλαια 3 και 4. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Φερνάντες ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί ένα ποσό δισεκατομμυρίων στο 1α, ωστόσο δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορώ να αποκλείσω να παρουσιαστούν σοβαρές ανάγκες λόγω της μετανάστευσης, ας πούμε, που μπορεί να χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν ώστε τις αρχές του 2020. Ε, ε, είναι μεγάλο πλεονέκτημα της ενδιάμεσης αναθεώρησης σε αυτή τη φάση. Υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξία ε, όμω και πρέπει να υπάρχει σε ένα τόσο άκαπτο προπολογισμό. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Είναι δύσκολο να βρεθεί ευελιξία σε έναν προπολογισμό που είναι τόσο άκαμπτο. Πώ θα αντιμετωπίσουμε καταστάσει κρίση. Το είδαμε το 2015 και το 2016. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω με τις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις. Νομίζω η επόμενη ερώτηση του κυρίου Φερνάντες ήταν ε, κατά πόσον αυτή η επαναχρησιμοποίηση θα προέρχεται από δωρεές ή από χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα προέρχεται και στις δύο περιπτώσεις από το ΣΕΦ Ενέργειας και το ΣΕΦ ICT από τις δωρεές. Σας το επιβεβαιώνω αυτό, είναι ξεκάθαρο. Και παρεπιπτόντω να πω ότι για το σεφ ενέργεια τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν υπάρχουν πλέον. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μετά την πρόταση τη χρηματοδότηση. Τέλο πάντων, ε, θεωρητικά. Διότι η πρόταση για το ΕΦΣΙ2 δεν έχει ακόμη εγκριθεί πλήρω. Αλλά η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να μην μείνει τίποτα. Η τελευταία ερώτηση του κυρίου Φερνάντε ήταν οι συνεισφορέ των κρατών μελών. Κατά τη δική μου κατανόηση, αυτά δεν θα περάσουν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, θα πάνε απευθεία ε, στον κλάδο. Ίσως όμω ο συνάδελφος ότι δίδει Γκρό μπορεί κάπω να βοηθήσει. Η τελευταία ερώτηση που σημείωσα είναι κατά πόσο η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον γεγονός ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην περίπτωση αυτή το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας παραπέμψω σε αυτό που είπε ο Επίτροπός μου, ο κύριος ήδη, σε αρκετές περιστάσεις, ότι δηλαδή ανησυχεί πολύ για την ύπαρξη χρηματοδοτικού χάσματος, το οποίο δημιουργείται από τη μια από το γεγονό ότι δεν θα συμβάλλει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο και από την άλλη από το γεγονό ότι θα υπάρξουν νέε ανάγκε για χρηματοδότηση. Και μεταξύ αυτών των νέων αναγκών για χρηματοδότηση είναι σαφέ ότι ο κύριος Έτιγκερ ε, τοποθετεί και τις ανάγκες χρηματοδότησης της άμυνας. Η άμυνα λοιπόν θα εντάσσεται σε αυτό το χάσμα χρηματοδότησης που έχει αναφέρει επανειλημμένος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου. Σας ευχαριστώ. Κάποια συνοπτικά σχόλια για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είπατε, πρόκειται για μια καινοτομία στον τομέα της βιομηχανίας της αμυντικής και της έρευνας. Είναι η λογική συνέπεια της προπαρασκευαστικής δράσης, η οποία είχε ξεκινήσει το 2016. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνέχιση δηλαδή της προπαρασκευαστικής αυτής δράσης και δεν τερματίζει την δραστηριότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπογραμμίσω ότι η πρόταση την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μια πρόταση για την πολιτική της άμυνας αλλά για την αμυντική βιομηχανία. Έχει σημασία η διαφοροποίηση. Το 173 είναι η νομική βάση, δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα. Είναι κάτι το οποίο άπτεται ε, του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας μάλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τώρα ποιος είναι ο στόχος της προτάσεώς μας. Εμείς διαπιστώσαμε πρώτον ότι υπάρχει μια έλλειψη συνεργασίας πολύ σημαντική στην Ευρώπη στον τομέα της βιομηχανίας της άμυνας της αμυντικής βιομηχανίας. Συγγνώμη. Υπάρχουν ε, σε κάθε κράτος μέλος ιδιαίτερα ανταγωνιστικές βιομηχανίες, αλλά το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσά τους είναι πάρα πολύ χαμηλό και αυτό δημιουργεί, ε, θα έλεγα, ένα επιπλέον κόστος για τον φορολογούμενο και μια καθυστέρηση ε, στην διαμόρφωση των δυνατοτήτων των στρατιωτικών τις οποίες έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Η προπασκευαστική δράση έχει σαν στόχο την άμυνα. Ο στόχος δεν είναι να μένουμε στην άμυνα, το θέμα είναι να εμπλουτίσουμε τις στρατιωτικές μας δυνατότητες. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία σε μια πρώτη φάση να προσκαλέσουμε με ευγένεια τις βιομηχανίες να συνεργαστούν αλλά αυτό δημιουργεί στην αρχή κάποιο επιπλέον κόστος. Ε, εκ των υστέρων θα υπάρξουν κέρδη σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Για να καλυφθεί το κόστος αυτό προτείνουμε τη συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή παίρνουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αλυσίδας των στρατιωτικών δυνατοτήτων, έχουμε καλύψει την έρευνα, πηγαίνουμε στην ανάπτυξη λοιπόν των μέσων τα οποία είναι καρπή της έρευνας. Δυστυχώς η έρευνα πολλές φορές δεν οδηγεί στην ανάπτυξη στη συνέχεια στον τομέα αυτό. Συνεισφέρουμε λοιπόν μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού με περιορισμένο τρόπο, καλύπτοντας το 20% του κόστους της ανάπτυξης των όπλων αυτών αλλά η συνεισφορά αυτή δεν είναι προβλέψιμη παρά μόνο σε επίπεδο συνεργασίας. Αν η βιομηχανία μας κάνει μια εθνική πρόταση, σαν παράδειγμα, δεν πρόκειται να το στηρίξουμε εφόσον είναι αυστηρά εθνικό. Εμείς θα στηρίξουμε μόνο τα διεθνή κοινοτικά προγράμματα με τρεις επιχειρήσεις κατελάχιστον και με δύο κράτη-μέλη επίσης κατελάχιστον. Στόχος είναι λοιπόν εμείς να ενισχύσουμε τις δυνατότητες αυτές της συνεργασίας. Προφανώς και υπάρχει εδώ κάποιο κόστος. Αν θέλουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της ανάπτυξης και μιλάμε για ένα προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων σε διετή βάση, το κόστος της ανάπτυξης είναι υψηλό, η άμυνα κοστίζει. Αν θέλουμε λοιπόν να διαφοροποιήσουμε κάπως την κατάσταση, φτάνουμε στα 500 εκατομμύρια. Αν καλύψουμε λοιπόν το 20% εμείς, το 80% θα πρέπει να το καλύψουν τα Υπουργεία Άμυνας που θα εμπλακούν στο συγκεκριμένο τομέα. Για να αποφύγουμε όμως να πάνε χαμένα τα χρήματα αυτά, προτείνουμε να υπάρξουν κάποιες προβλέψεις οι οποίες να ε, ζητούν από τα κονσόρτιουμ των επιχειρήσεων να αποδεικνύουν ότι έχουν ήδη ε, την σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών να διασφαλίσουν ε, να χρησιμο, την χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας. Με λίγα λόγια να μην παράγουμε προϊόντα τα οποία θα μείνουν στο ράφι και τα οποία κανένας δεν θα χρησιμοποιήσει εκ των υστέρων. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, εδώ βρισκόμαστε στην παρούσα φάση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν, υπάρχει ακόμα μια κάποια ρευστότητα πολιτική ε, για τον τομέα της άμυνας ε, ε, η κυρία Γκρέσλερ. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις. Η ερώτηση παραμένει ένας διαγωνισμό για αμυντικά όπλα ή για αμυντικά προϊόντα μπορώ να, την να τον οργανώσω εγώ ανεξάρτητα από το τι ε, αποφάσεις θέλω να πάρω και τι προϊόντα θέλω να αγοράσω. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προέλθει αυτό από το 20% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Αυτό δεν το θέλω. Ότι χρειαζόμαστε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την αμυντική βιομηχανία. Ναι, φυσικά, αλλά νομίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε. Να το ξαναδούμε και να καλέσουμε ίσω ε, και του ανώτερου να φέρουμε εδώ τον Επίτροπο Έτινγκερ, γιατί είναι ένα θέμα ουσιώδε. Και στην τελευταία συνάντηση ε, για τον προπολογισμό είχαμε πει 25 εκατομμύρια για τέτοια πιλωτικά προγράμματα και εκεί είχα πει ότι είναι το πρώτο λάθος. Τώρα είμαστε ε, έτοιμοι να κάνουμε το δεύτερο λάθος. Δεν πρέπει να χάσουμε τη γενική δομή, τη γενική αρχιτεκτονική του συστήματος. Και δεν θέλω τώρα να πω ότι ικανοποιήθηκα από αυτά τα μικρά ψήγματα που μας έδωσε η Κομισιόν. Για ένα τέτοιο θέμα λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι καλό να στέλνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο στόμα του λύκου τους απλούς υπαλλήλους. Καλό θα ήταν να έρθουν εδώ τα μεγάλα κεφάλια και να μας δώσουν τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε θα πρέπει εδώ να συμφωνήσω με την κυρία Γκρέσλε. Από την πλευρά της Ευρώπης πολιτικώς τι θέλουμε. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί. Διότι έχουμε την εντύπωση ότι βάζουμε κομματάκια ζάχαρης ε, στη διαδρομή, ελπίζοντας ότι τα πάει ο κόσμο να τα αρπάξει. Αλλά βλέποντα τι επιφυλάξεις των μεγάλων κρατών, σε εθνικό επίπεδο και των ε, επιχειρηματιών, που βεβαίως είναι σε άμεση συνεργασία με τα γενικά επιτελεία, ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτικό εγχείρημα, πολιτικό όραμα που να το στηρίζει η κοινή γνώμη και να έχει πολιτική αξία. Ε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από μαστορέματα, πρόχειρες και προσωρινές λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε ότι θα είμαστε πολύ μετριοπαθείς στην προσέγγιση μας και θα είναι συμβολική η προσφορά μας. Πρέπει να δοθεί μια νέα ευρωπαϊκή πνοή σε όλα αυτά, Όπως είπε και ο κ. Κέλμεν. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει προσταθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή συμβολή. Ποια είναι αυτά τα δημόσια αγαθά που μόνο η Ευρώπη μπορεί να διασφαλίσει για τους πολίτες μας αύριο, στο μέλλον. Ποιοι είναι αυτοί που σε εθνικό επίπεδο μπορούν να τα διασφαλίσουν και τη στιγμή της παγκοσμιοποίησης τι είναι αυτό που θα πρέπει να αναλάβει το ευρωπαϊκό επίπεδο αφού το εθνικό δεν μπορεί πια να το καλύψει. Ίσως τέλο πάντων ε, να παραμένουμε σε αυτά σήμερα. Ήταν μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, ε, η οποία όμως μας ε, προχωρεί και μας φέρνει σε άλλες πολιτικές συζητήσεις και σε μια συνέχεια. Θα διακόψουμε συνάδελφοι τις εργασίες μας για να ξαναρχίσουμε στις τρεις. Τρεις με το ρολόι, έτσι. Oui, ben on dira να διευκρινίσω ότι στι 3 είναι και κλεισμένο των θυρών η συνεδρίαση. Για κάποιου από εσά ε, διοργανωθείτε αναλόγω. C'est pas vous déranger.